Good morning. Good morning, Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Μου λέγουν ότι μπορούμε να αρχίσουμε, γιατί είναι και ο συνάδελφος Λάγκ εδώ πλέον μαζί μας. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχουν παρατηρήσεις για την ημερήσια διάταξη, δεν βλέπω. Ανακοινώσει του Προέδρου. Δεν έχω τίποτα να σας πω. Έγκριση των πρακτικών που υπάρχουν online 11 Ιανουαρίου, 28 Ιανουαρίου, 22, 23 Φεβρουαρίου. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, θα θεωρηθούν ότι εγκρίθηκαν τα πρακτικά. Ε, ευχαριστώ πολύ. Σημείο 4 στην ημερήσια διάταξη συζήτηση για το καθεστώς οικονομίας της αγοράς στην Κίνα ενδεχόμενες συνέπειες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η παρουσίαση θα γίνει από τον Διευθυντή Λεοπόλντο Ρουμπινάτσι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλώς ήρθατε Διευθυντά. Να καλωσορίσω και τον συνάδελφο Μπέρντ Λάνε που είναι ο υπεύθυνος για το Διεθνές Εμπόριο ως ε, πρόεδρο της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ. Μια σύντομη εισαγωγή. Η Κίνα προσχώρησε στον ΠΟΕ το 2001. Οι διαπραγματεύσεις ε, ασχολήθηκαν με το πώς τα μέλη του ΠΟΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να χορηγήσουν ε, καθεστώς οικονομίας της αγοράς στην Κίνα σε ένα μεταγενέστερο στάδιο. Αυτές ήταν οι διαπραγματεύσεις στην αρχή, όταν προσχώρησε δηλαδή η Κίνα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Το καθεστώς της οικονομίας της αγοράς έχει άμεση επίπτωση στις βιομηχανίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να προστατεύσει την οικονομία της από αθέμητες πρακτικές όπως dumping, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και άλλες μορφές dumping και θέλουμε να δούμε πώς η Κομισιόν σκέφτεται να αντιμετωπίσει το θέμα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση σκέπτεται να χορηγήσει αυτό το καθεστώς στην Κίνα τώρα, ε, σε αυτή τη ε, φάση γιατί μας εξέπλησε λίγο γνωρίζοντας την ε, κατάσταση της οικονομίας αγοράς στην Κίνα. Δεύτερη σημαντική ερώτηση. Ο αντίκτυπος που θα έχει η χορήγηση του καθεστώτος στην Κίνα στις βιομηχανίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ολόκληρη η ευρωπαϊκή οικονομία θα έχει επιπτώσεις, κυρίως η βιομηχανία όμως ίσως δεν ενδιαφέρεστε τόσο πολύ, δεν, ενδια... είναι τόσο ενδιαφέρον το θέμα της γεωργίας εδώ, αλλά και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εμείς θα συζητήσουμε για τις βιομηχανίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ίσως και θέματα ενέργειας. Αλλά και ένα τρίτο ερώτημα υπάρχει. Τα άλλα μέλη του ΠΟΕ, όπως οι Ηνωμένε Πολιτείες, πώς αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό. Γιατί βεβαίως ε, θέλουμε ενδεχομένως να έχουμε ένα κοινό μέτωπο και με άλλους. Είναι σημαντικό αυτό προκειμένου περί της παγκόσμιας οικονομίας της αγοράς. Κύριε Διευθυντά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτό το θέμα στην Επιτροπή σας. Έχετε δίκιο κύριε Πρόεδρε ότι είναι θέμα εμπορικό αυτό, αλλά έχει σημαντική επίπτωση στη βιομηχανία. Καταρχήν, να ορίσω το θέμα μας. Περί τίνος ομιλούμε. Δεν ομιλούμε για την απόφαση ενδεχομένως αν είναι ή δεν είναι η οικονομία της αγοράς η Κίνα. Ποιοι είμαστε εμείς για να πάρουμε μια τέτοια απόφαση. Πρέπει να αποφασίσουμε αν και αν θα το κάνουμε πώς, πρέπει να αλλάξουμε την νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με τη μέθοδο με την οποία υπολογίζουμε το dumping ε, στις έρευνες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το αντι-dumping. Δεν το λέω αυτό για να υποβαθμίσω τη σημασία του θέματος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Το λέω για δύο λόγους. Πρώτον, νομίζω ότι είναι σημαντικό να είμαστε πολύ ακριβείς Δεύτερον, επειδή το θέμα του καθεστώτος είναι διτό θέμα. Είτε έχουμε, είτε, ε, ε, δεν είναι διτό, έχουμε είτε δεν έχουμε ε, καθεστώς. Το θέμα της μεθοδολογίας είναι ένα άλλο θέμα. Πώς θα βρούμε λύση δηλαδή. Όπως λέτε, όταν προσχώρησε στον ΠΟΕ το 2001 η Κίνα, υπήρχε ένα πρωτόκολλο το οποίο το διαπραγματεύτηκαν και έθετε συγκεκριμένους κανόνες σε σχέση με την Κίνα. Και ένας από αυτούς τους κανόνες ασχολείται με τη μέθοδο με την οποία τα άλλα μέλη του ΠΟΕ μπορούν να υπολογίσουν το dumping στις έρευνες αντι-dumping για την Κίνα, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Κίνα σε αυτή τη φάση, τότε το 2001 δηλαδή, αλλά και ακόμα και σήμερα θα έλεγα, δεν ήταν η οικονομία της αγοράς, άρα το dumping ήταν ε, ε, ε, ως σύγκριση τιμών υπολογίζεται, υπολογίζοντας τις τιμές ενός προϊόντος στην εγχώρια αγορά της Κίνας και συγκρίνονται με τις τιμές του ιδίου προϊόντος όταν εξάγεται στην Ένωση, δηλαδή η τιμή από την Κίνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι οι τιμές που τίθενται από την αγορά, γιατί η αγορά αποφασίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εγχώριε τιμέ στην Κίνα ω επιτοπλίστων δεν καθορίζονται από την αγορά. Το βασικό πρόβλημα λοιπόν στον υπολογισμό του ντάμπινγκ είναι πώ συγκρίνονται αυτέ οι τιμέ. Και επειδή η Κίνα δεν είναι η οικονομία της αγοράς, το πρωτόκολλο της προσχώρησης της Κίνας ανέφερε ε, κάποιες εναλλακτικές, εκτός από την ε, παραδοσιακή, δηλαδή την άμεση σύγκριση των τιμών. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι κάποιες διατάξεις του πρωτοκόλλου αυτού λήγουν στις 11 Δεκεμβρίου τρέχοντος. Οπότε η απάντηση στο ερώτημά σας γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση το εξετάζει το θέμα τώρα, ε, το εξετάζει διότι υπάρχει προθεσμία καταληκτική. Γιατί δεν το εξέτασε προηγουμένως. Το εξέτασε η Ευρωπαϊκή Ένωση και παλιότερα το θέμα αυτό και κάποια στιγμή οι επίτροποι θεώρησαν ότι το θέμα είναι τόσο σημαντικό ώστε πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης θεώρησε ότι θα έπρεπε να υπάρχει πλήρης εξέταση των ενδεχομένων επιπτώσεων. Γι' αυτό τώρα διεξάγει μια εκτίμηση επιπτώσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί διαφόρων εναλλακτικών αντιμετώπιση του θέματος. Το θεμελιώδες ζήτημα είναι αν και πώς θα γίνει η τροποποίηση της νομοθεσίας, αν αυτή χρειάζεται. Υπάρχουν τρεις εναλλακτικέ. Η πρώτη να μην κάνουμε τίποτα. Η δεύτερη είναι να αντιμετωπίσουμε την Κίνα με την παραδοσιακή νομοθεσία, ε, μεθοδολογία όπως την Νότια Κορέα για παράδειγμα και η τρίτη εναλλακτική είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε μια εναλλακτική μέθοδο η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις τρευλώσεις που υπάρχουν στην κινέζικη αγορά ώστε να εφόσον η μέθοδος αυτή θεσμοθετηθεί, να συνεχίσουμε να μπορούμε αποτελεσματικά να αντιμετωπίζουμε τις πρακτικές dumping από την Κίνα. Παρά την ε, εκτίμηση επιπτώσεων κάνουμε και δημόσια διαβούλευση που τελειώνει στις 20 Απριλίου. Είχαμε μια πολύ επιτυχημένη συνάντηση με τους Ευρωπαίους εμπλεκομένους το προηγούμενο μήνα περίπου 300 εμπλεκόμενοι από διάφορους τομείς, έμποροι, εξαγωγή, παραγωγή κλπ. Και με την παρουσία της Επιτρόπου Μάλμστρομ είχαμε μια καλή συζήτηση και θα έχουμε και με τους κοινωνικούς εταίρους της Ένωσης συνάντηση. Κάνουμε ευρύτατες διαβουλεύσεις. Οι Επιτροποί αποφάσισαν να επανέλθουν στο θέμα αυτό στις 13 Ιουλίου. Οπότε δεν θα ακούσετε τίποτα συγκεκριμένο από την Επιτροπή πριν από τις 13 Ιουλίου. Λοιπόν, υπάρχουν επιπτώσεις. Ποιες είναι στη βιομηχανία. Πρέπει να πω από την αρχή ότι ο υπολογισμός του αντίκτυπου είναι πολύ δύσκολος. Γιατί. Ο βασικός λόγος είναι ότι οι έρευνες αντι-dumping είναι ε, πάνω στη βάση της συμμόρφωσης. Με την έννοια ότι πριν αρχίσουμε μία έρευνα πρέπει να υπάρξει καταγγελία από ένα κλάδο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Σήμερα δεν ξέρω τι καταγγελίες και παράπονα θα λάβουμε μέσα σε δύο μήνες ή μέσα στον επόμενο μήνα. Οπότε δεν μπορώ να σας πω και τι είδους έρευνες πρόκειται να χειριστεί η Κομισιόν. Ο δεύτερος θεμελιώδης λόγος ε, ε όπου υπάρχει πρόβλημα είναι ότι η, ποσότητα, ο όγκος του ντάμπινγκ είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένου υπολογισμού που λαμβάνει υπόψη τις καθ' αυτό συναλλαγές, τις πωλήσει που λαμβάνουν χώρα ε, στα πλαίσια του εμπορίου ε, ε, Κίνας. Οπότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε υποθέσεις, να δουλέψουμε με βάση υποθέσεις εργασίας. Κάναμε έπανα υπολογισμούς παλιών υποθέσεων για να δούμε τι περιθώρια dumping έχουμε. Κάναμε ένα πρώτο υπολογισμό που βλέπει τι θα γινόταν αν θα αντιμετωπίζαμε την Κίνα ακριβώς όπως αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε οικονομία της αγοράς στον κόσμο, Νότια Κορέα ή Ηνωμένε Πολιτείε, για παράδειγμα. Και βλέπουμε ότι το πραγματικό επίπεδο των δασμών αντι-dumping που θα μπορέσουμε να επιβάλλουμε θα είναι χαμηλότερο κατά περίπου 27%. Οπότε ε, είναι στατιστικά σημαντική μείωση. Και υπολογίσαμε ότι η, η δυνητική επίπτωση σε ό,τι αφορά θέσεις εργασίας στη βιομηχανία και αυτό μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή μιλάμε για 200 250000 χιλιάδες ε, θέσεις στη βιομηχανία, θέσεις εργασίας στη βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θα μπορούν πλέον να προστατεύονται από ε, δυνητικά μέτρα αντι-dumping. Οπότε και εδώ είναι ενδεχομένως σημαντικός ο αντίκτυπος. Δεν έχουμε τελειώσει του υπολογισμού, γιατί θέλουμε να υπολογίσουμε και το τι θα συμβεί αν επρόκειτο να εφαρμόσουμε εναλλακτική μεθοδολογία. Ο πυρήνα τη εναλλακτική, που είναι η εναλλακτική τρία στην ε, μελέτη επιπτώσεων, είναι μια μεθοδολογία που θα μα επέτρεπε, όπω κάνουμε σήμερα, αλλά με άλλα μέσα, με άλλου τρόπου, να μην λάβουμε υπόψη μα το κόστο παραγωγή τη Κίνα, να το αφαιρέσουμε όταν υπολογίζουμε το dumping. Γιατί για να έχουμε ε, ένα υποκατάστατο αυτών των τιμών και του κόστους που δεν επηρεάζεται από τις πολλές τρευλώσεις στην κινέζικη αγορά. Τώρα πάμε να τελειώσουμε τους υπολογισμούς που προφανώς θα συμπεριληφθούν στην ε, μελέτη επιπτώσεων και μετά υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία ε, της εναλλακτική μεθοδολογίας που ευχαρίστως να σας τα πω αν ερωτηθώ σχετικά. Ο αντίκτυπος λοιπόν, οι επιπτώσεις, αν πάμε προς ολοταχώς προς μια αντιμετώπιση της Κίνας ως οικονομία της αγοράς μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντική για τις, νέα, για τις θέσεις εργασίας. Οι επιπτώσει του να μην κάνουμε τίποτα επίσης θα είναι σημαντικές. Γιατί διότι αν και οι δικηγόροι διαφωνούν για την ακριβή σημασία του πρωτοκόλου, Υπάρχει μια παράγραφο στο πρωτόκολλο που λίγη δεν θα υφίσταται ούτω ή άλλω. Και η λήξη αυτή τη παραγράφου στο πρωτόκολλο που θα γίνει ούτως ή άλλως μπορεί νομικά να σημαίνει ότι η αλλω μπορει μέθοδος που χρησιμοποιεί η τωρινη μέθοδο που Ένωση μπορεί να μην συνάδει με τον ΠΟΕ. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μόνος μεγάλος χρήστης, ε, χρήστης που έχει δύο στοιχεία στην νομοθεσία του. Το πρώτο είναι σαφής ε, αναφορά στην Κίνα, αναφέρεται ρητά στην νομοθεσία μας. Η Κίνα και δεύτερον υπάρχει μια υποχρέωση όταν γίνονται έρευνες για την Κίνα σε σχέση με το αντι-dumping να χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένη μέθοδος που λέγεται η μέθοδος της ανάλογης χώρας. Είναι μια μέθοδος με την οποία υποχρεούμεθα να χρησιμοποιήσουμε τιμές ή κόστη σε μια τρίτη χώρα, όχι την Κίνα, όταν υπολογίζουμε το ντάμπινγκ. Αυτό δημιουργεί μια ιδιαιτερότητα για την Ένωση. Οι ΗΠΑ δεν έχουν το ίδιο σύστημα. Έχουν άλλο σύστημα οι Ηνωμένε Πολιτείε, όπου καταρχήν το Υπουργείο Εμπορίου έχει, κάνει ε, μια, έχει πάρει μια απόφαση ότι δεν είναι οικονομία της αγοράς, αυτό είναι κατατεθειμένο και επί τη βάση αυτής της απόφασης οι ε, ερευνητικέ αρχές των ΕΠΑ έχουν ε, μια γκάμα εναλλακτικών μεθοδολογιών. Σήμερα οι Αμερικανοί λοιπόν δεν είναι στην ίδια θέση με εμάς. Και προσθέτω ότι ενώ εμείς πρέπει να αλλάξουμε την νομοθεσία μας, αν αποφασίσουμε ότι κάτι πρέπει να γίνει, οι Αμερικανοί και οι Ιάπωνες και οι Καναδοί ακόμα μπορεί να κάνουν τροποποιήσεις με βάση διοικητική απόφαση και μόνο. Οπότε έχουμε πολλές επαφές με τους συναδέλφους μας σε άλλες σημαντικές χώρες, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι έχουμε μια ιδιαίτερη και ειδική θέση που σημαίνει ότι μειώνεται σε ένα βαθμό η δυνατότητα συντονισμένης δράσης, δηλαδή συγχρονισμένης δράσης. Σταματώ εδώ, μια και μου φαίνεται ότι μίλησα πολύ, αλλά ε, θα είμαι ευτυχής να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά για τις εξηγήσεις και τις παρατηρήσεις σας. Ο, δίνω το λόγο στον κύριο Λάγκε καταρχήν, ε, πρόεδρο της Επιτροπής Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που με καλέσατε ως Πρόεδρο της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ. Η Κίνα πράγματι αποτελεί πρόβλημα σε σχέση με το dumping και παράνομες επιδοτήσεις. 80% περίπου των περιπτώσεων που μας απασχολούν σχετίζονται με την Κίνα. Οπότε η ερώτηση του τι θα γίνει μετά τις 11 Δεκεμβρίου ε, είναι πολύ σημαντική. 11 Δεκεμβρίου υπενθυμίζω ότι ε, λύγει το πρωτόκολλο ε, ένταξη της ε, Κίνας στον ΠΟΕ. Έχουμε το παράδειγμα της Αυστραλίας στο παρελθόν όπου αριθμός, ο αριθμός των περιπτώσεων που, ε, των καταγγελιών ε, μειώθηκαν στο μισό μειώθηκε στο μισό. Μόνο, το 50%, μόνο για το 50% των περιπτώσεων ε, βρέθη, ε, μπόρεσαν να ε, διερευνηθούν και οι δεσμοι αντιντάπινγκ αντι-dumping μειώθηκαν στο 10%, το οποίο είναι μηδενικό σχεδόν. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το σύστημά μας να μας εγγυάται ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να αντιδράσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις ε, dumping και ε, παράνομων επιδοτήσεων. Για παράδειγμα, στο Χάλιβα, όπως επίσης στο, μέλλον θα, σύντομα θα έχουμε και πολλά προβλήματα με τις ανεμογεννήτριες. Ε, η αγορά κατακλείζεται από κινέζικα προϊόντα, 33% αυτή τη στιγμή το μερίδιο της Κίνας. Ε, μια αύξηση δηλαδή άνω του 50% σε ένα χρόνο. Έχουμε προϊόντα dumping ε, ε, από την Κίνα σε μεγάλο βαθμό και σε μεγάλους αριθμούς. Θα πρέπει να προστατευτούμε. Οπότε έχουμε δύο προβλήματα. Πρώτον, τα μέσα που διαθέτουμε για την εμπορική άμυνα είναι πεπαλαιωμένα. Θα πρέπει να τα ανανεώσουμε. Ως Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2014 υιοθετήσαμε ένα πακέτο εξυγχρονισμού που δίνει στην Κομισιόν την ευελιξία να ξεκινάει ε, έρευνες ε, όχι μόνο κατόπιν καταγγελιών αλλά αυτεπάγγελτα. Όμως το Συμβούλιο από τον Απρίλιο του 2014 μπλοκάρει αυτόν τον εξυγχρονισμό και έχουμε ε, κινητοποιηθεί προκειμένου το Συμβούλιο να το υιοθετήσει αυτό το πακέτο, να έχουμε ένα πραγματικό, μοντέρνο, σύγχρονο σύστημα anti-dumping. Και δεύτερον, χρειάζεται να μεταρρυθμίσουμε το δικό μας σύστημα σε σχέση με την Κίνα, έτσι ώστε να διαθέτουμε επαρκείς μηχανισμούς μετά, την 11η Δεκεμβρίου. Πρότασή μας είναι μια εναλλακτική μέθοδος υπολογισμού του dumping και της κατάχρησης επιδοτήσεων μετά την 11η Δεκεμβρίου. Οπότε ζητούμε από την Κομισιόν να υποβάλει ένα, μια πρόταση. Είχε 15 χρόνια να το σκεφτεί. Ελπίζω ότι μια τέτοια πρόταση θα υποβληθεί σύντομα. Η Επιτροπή Ίντα θα υιοθετήσει στην Ολομέλεια του Μαΐου ένα ψήφισμα σχετικό. Ευχαριστώ. Κυρία Αγγέλικα Νίβλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον εκπρόσωπο της Κομισιόν για τις ε, παρατηρήσεις του. Να κάνω μερικές παρατηρήσεις και μία ερώτηση. Τα εμπορικά θέματα δεν τα γνωρίζω τόσο καλά όσο ο συνάδελφος Λάνε. Λοιπόν, επιτρέψτε μου κάποιες παρατηρήσεις. Είπατε ότι δεν είναι μόνο εμπορικό το θέμα, αλλά το καθεστώς ε, οικονομίας της αγοράς ε, της Κίνας είναι και θέμα βιομηχανικής πολιτικής. Η ομάδα μας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη ε, στη συζήτηση που γίνεται γιατί έχει μεγάλη πολιτική σημασία και ανησυχούμε κιόλας ότι ένα κομμάτι της βιομηχανικής μας παραγωγής θα φύγει από την Ευρώπη αν ληφθούν οι λάθος αποφάσεις. Τονίζω ότι δεν πρόκειται για προστατευτισμό εδώ, γιατί αυτό, γι' αυτό μας επικρίνουν οι Κινέζοι. Το θέμα είναι να υπάρχει δίκαιος ανταγωνισμός. Και πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Πρόκειται για δικαιότερες συνθήκες ανταγωνισμού. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σχετικά με το χειρισμό του θέματος φέτος και βεβαίως σε σχέση με τη χορήγηση του καθεστώτος οικονομίας της αγοράς στην Κίνα. Ερώτηση λοιπόν προς εσάς γιατί το συσχετίσατε το θέμα και με τη νέα εκδοχή, τροποποίηση της νομοθεσίας, αλλαγή της, νομο... μεθοδολογίας και προσθέσατε ότι στις Ηνωμένε Πολιτείες το σύστημα είναι διαφορετικό. Η διοίκηση δηλαδή κινείται διαφορετικά και έχει άλλα περιθώρια ευελιξίας μεγαλύτερα. Ρωτώ λοιπόν λίγο ομά, γιατί δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε κι εμείς το σύστημα των Αμερικανών ούτως ώστε να κάνουμε τη δουλειά μας ευκολότερη. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Μιλήσατε και για την εκτίμηση επιπτώσεων που είναι τώρα υπό προετοιμασία. Αυτή η εκτίμηση επιπτώσεων πότε θα είναι διαθέσιμη, πότε θα κυκλοφορήσει, ούτω ώστε να έχουμε αρκετό χρόνο να την λάβουμε υπόψη μας. Ε, μιλήσατε για τρεις αναλλακτικέ. Εγώ τις συζητήσεις εδώ δεν τις παρακολουθώ εκ του σύνεγγης, αλλά αναφέρατε τις τρεις μεθοδολογίες, και ρωτώ, θα μπορούσε να υπάρξει και μια τέταρτη εναλλακτική, εκτός από τις τρεις αυτές που αναφέρατε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Νίμπλερ ε, από το ΕΛΚ. Η κυρία Κάρτον Ντάρλινγκ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Θα είμαι σαφής. Αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, περνάμε από μια επαξιακή κρίση στην βιομηχανία ε, του Χάλιβα. Ε, 48.000 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή ε, περιμένουν να δουν πώς θα γίνει, ποια θα είναι η τύχη τους και αν θα πουληθεί η βιομηχανία Χάλιβα του Ηνωμένου Βασιλείου. Όλα αυτά έχουν σχέση με το, με το μαζικό dumping προϊόντων από την Κίνα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Και όλα αυτά δυσχεραίνονται από το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο έκανε τη δουλειά του προσπαθώντας να ενισχύσει τους αμυντικούς μηχανισμούς της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά το, η κυβέρνησή μας στο Συμβούλιο των Υπουργών είναι, ε, αποτελεί ε, το πρόσκομα το οποίο μπλοκάρει την υιοθέτηση αυτού του μηχανισμού που θα προστάτευε τη βιομηχανία μας. Οπότε επικρατεί μια πραγματική πικρία στον Βασίλειο για την κατάσταση. Τώρα γίνεται μια σύγχυση ανάμεσα στους μηχανισμούς εμπορικής άμυνας που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή στο επόμενο Συμβούλιο Εμπορίου στις 15 Μαΐου και εκεί οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ξεμπλοκάρουν το θέμα αυτό η Ιταλική Προεδρία ήδη έχει υποβάλει προτάσεις, μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα για να βρούμε ένα συμβασμό στο Συμβούλιο. Αυτό πρέπει να γίνει αφενός. Ε, οι κυβερνήσεις μας από την άλλη μεριά πρέπει να μιλήσουμε με την κυβέρνηση της Κίνας προκειμένου να δούμε τι θα γίνει με το θέμα της, ε, ε, του υπερβάλλοντος δυναμικού στην οικονομία της Κίνας. Ε, από την άλλη μεριά, από τη δική σας μεριά περιμέναμε 15 χρόνια, εντάξει ήταν πολύ, παρόλα αυτά δεν μπορούμε να ξαναγράψουμε την ιστορία. Ε, τι γίνεται αυτή τη στιγμή από πλευρά διαλόγου μεταξύ κομισιών και άλλων χωρών του ΠΟΕ που θα πρέπει να πάρουν απόφαση. Ε, στις ΗΠΑ είναι τεχνική πιο πολύ απόφαση, αλλά για τη Βραζιλία, τον Καναδά και άλλες χώρες η απόφαση δεν είναι τεχνική. Συντονίζεστε με αυτού. Μπορείτε να παρουσιάσετε ένα ενιαίο μέτωπο έτσι ώστε η απόφαση να είναι κοινή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έριξον Γκριντς. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που υπόθηκαν. Κύριε Ρουμπινάτση, μια ερώτηση. Μιλάμε για την Κίνα. Δεν είναι μια οικονομία της αγοράς 100%. Όλοι το ξέρουμε. Υπάρχουν δύο προβλήματα. Μάλιστα. Κάτι που ξέρουμε εδώ και καιρό, ότι δεν είναι μία 100% οικονομία της αγοράς η Κίνα. Και κάτι άλλο όμως που υπόθηκε, ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα τεράστιο πλεονάσμα δυναμικό στην παραγωγή της Κίνας, παράδειγμα το χάρη χάλιβα. Η παραγωγή του χάλιβα είναι τεράστια. Και αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ακόμα και σε μια οικονομία τη αγορά, όταν έχει τεράστια παραγωγή, οι τιμέ ε, πέφτουν και πολύ κάτω από το κόστο παραγωγή συχνά. Το είδαμε, παραδείγματο χάρη, στο πετρέλαιο. Κατα, ε, οι τιμέ. Γιατί έχουμε τεράστιο δυναμικό παραγωγή. Πολύ μεγαλύτερο από την κατανάλωση. Τι θα κάνει η Κομισιόν για αυτό το πλεονάσμα δυναμικό τη μείωση των τιμών, πολύ κάτω από το κόστος παραγωγής. Τα λαμβάνετε αυτά υπόψη σας στην ανάλυση σας, Κομισιόν. Κύριε Λόπες Μπερμέο, από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Διευθυντή. Σε αυτή τη φάση είναι σαφές ότι το καθεστώς αυτό στην Κίνα ε, θα πλήξει πολλούς τομείς που είναι σε κρίση. Παραδείγματος χάρη η κεραμική, ε, ή η βιομηχανία ε, εξαρτημάτων ε, για τα αυτοκίνητα, παραδείγματο χάρη. Επίσης, η σιδηρουργία. Γιατί όπως αναγνωρίστηκε από τον Αντιπρόεδρο Κατάινεν εδώ στην Επιτροπή μας και από την ανακοίνωση της Επιτροπής, πρόκειται για ένα τομέα στην κρίση σε όλη την Ευρώπη. Και υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες για ντάμπινγκ που τρέχουν. Έχει σχολιαστεί αυτό. Γι' αυτό η θέση μας είναι αντίθετη στο να δοθεί το καθεστώς οικονομία αγοράς στην Κίνα. Ε, υπάρχει αντική επίπτωση στην απασχόληση. Μία ε, μελέτη μιλάει για τις απώλειες ότι θα είναι 1,7 με 3,5 εκατομμύρια απώλειες θέσεων εργασίας και με αυτά τα νούμερα τα λαμβάνετε υπόψη Λαμβάνεται υπόψη επίσης την απώλεια κοινωνικού ιστού. Ε, θα χάσουμε και τεχνολογικό δυναμικό, θα, χάσουμε, θα μειώθει και η ζήτηση και βεβαίως θα πέσουν και οι μισθοί και θα υπάρξει ανεργία. Τα λέω γιατί επίσημες μελέτες του TTP, παραδείγματος χάρη, χρησιμοποιούν την υπόθεση ότι θα υπάρχει αυτόματα πλήρης απασχόληση. Αυτό είναι εντελώς αναξιόπιστο δεδομένο στον άλλων, ε, των επιπτώσεων που είχαν άλλες συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Ε, έχετε διμερείς επαφές μέσω των οποίων ε, αποφασίζετε να επιταχύνετε την χορήγηση του καθεστώτος στην Κίνα. Δεν υπάρχει καμία εντολή για να παραταθεί επαορίστο η σημερινή κατάσταση. Τέλος, πιστεύουμε ότι η παραχώρηση του καθεστώτος αυτού θα πρέπει να λάβει υπόψη παράγοντες όπως τα κοινωνικά πρότυπα για τις, τις ε, συλλογικές ε, διαπραγματεύσεις. Η αγορά δεν είναι ένας φυσικός ε, θεσμός, ας πούμε. Δημιουργείται και εάν έχουμε μόνο, απελευθε... και, και όχι καθόλου κοινωνικά πρότυπα, αυτό θα ήταν πρόβλημα. Δεν θα ήθελα μέσω της απελευθέρωσης αυτής να ε, διαλύσετε ακόμα περισσότερο την αγορά εργασίας. Ο κ. Μπορέλη. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, αλλά ξεκινάω από τη θέση της ομάδας μου, που ήταν πάντα ξεκάθαρη. Δηλαδή, κανένα πρόβλημα κατά της συνεργασίας ε, και της εμπορικής συνεργασίας με την Κίνα δεν θα πρέπει να επιβληθεί λόγω του φόβου οτιδήποτε. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα ε, γεγονότα και στα συμβάντα και να λάβουμε υπόψη μας την νομοθεσία το Better Regulation. Επίσης, πέστε μου, πώς υπολογίσατε όλα αυτά που μας είπατε, γιατί τα νούμερα μας εκπλήσουν. Τα άλλα ε, ερωτήματά μας αφορούν την δημόσια διαβούλευση. Μας εντυπωσίασαν τα όρια που επιβλήθηκαν. Νομίζουμε ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Πρώτον, ε, όλα αυτά διατυπώνται με πάρα πολύ τεχνικό τρόπο και επομένω περιορίζεται προφανώ η συμμετοχή. Δεν μα επιτρέπει ανοιχτέ απαντήσει. Ε, μπλοκάρει την επιχειρηματολογία, είναι εντελώ ε, προσανατολισμένε και ξεκινάται από, την, ε, από το δεδομένο ότι είναι υποχρεωτικό να δοθεί αυτή, αυτό το καθεστώ οικονομία τη αγορά στην Κίνα. Γιατί αυτέ οι επιλογέ στη δημόσια διαβούλευση. Επίση, στη δημόσια στη δημόσια διαβούλευση. Πώς θα αξιολογήσετε ε, φορείς ή άτομα τα οποία δεν ε, διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το θέμα της ε, μελέτης αντικτύπου. Ποιος το κάνει. Και ακόμα και αν παρουσιαστεί αύριο το πρωί, πώς μπορούμε τόσο σύντομα να σας δώσουμε ε, απόψεις και εν πάση περιπτώσει πώς μπορείτε να δώσετε ε, αμυντικά εργαλεία στις επιχειρήσεις μια και η καταληκτική ημερομηνία είναι 11 Δεκεμβρίου. Με όλα αυτά τα δεδομένα που έχετε στην ε, διάθεσή σας, με βάση την εμπειρία σας λοιπά Κατά την άποψή σας τι θα συμβεί στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και σε εκείνους τομείς όπως το, ε, το ο Χάλιβας και ο κατασκευαστικός τομέας και τι θα γίνει κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τι θα γίνει με το μέγεθός τους. Θα αντέξουν. Έχω διάφορες ε, ερωτήσεις. Πρώτον, μια παλιά συζήτηση με τον ΠΟΕ, με τον Πασκάλ που δεν ε, θέλαν τότε να αναγνωρίσουν τα γεγονότα. Δηλαδή, ότι η απελευθέρωση των συναλλαγών οδηγεί σε μαζική καταστροφή ε, θέσεων εργασία στη βιομηχανία στην Ευρώπη. Στη χώρα μου, από τότε που είναι στην εξουσία οι σοσιαλιστές, από το 12% του ΑΕΠ ε, σε προστιθέμενη αξία, πήγαμε στο μισό. Αυτή η μαζική καταστροφή ε, θέσεων απασχόλησης στην βιομηχανία όχι μόνο θα πρέπει να, λάβουν, τις δούμε υπό την ε, έννοια της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας. Και αυτό είναι συζητήσιμο. Αλλά τι θα γίνει αν το, τις εξετάσουμε ε, σε σχέση με τις μακροπρόθεσμες ε, συναλλαγές. Η χάρτα της Αβάνας μετά τον πόλεμο πρότεινε ισορροπία των συναλλαγών για να υπάρχει βιώσιμο εμπόριο. Φυσικά δεν είναι κατά της Κίνας. Έχω και φίλους Κινέζους. Γνωρίζω την Κίνα, πήγα και εκπροσώπησα τα γαλλικά συμφέροντα στην Κίνα. Μιας γαλλικής δηλαδή εταιρεία. Αλλά θα πρέπει να δούμε τη σχέση μας μακροπρόθεσμα. Δεν μπορούμε να έχουμε πλεονάσματα από τη μία και μονίμω ελλείμματα από την άλλη. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να έχουμε συστηματική καταστροφή τη δική μα βιομηχανική βάση γιατί είναι θέμα κυριαρχίας μας, ανεξαρτησίας μας, αλλά και ικανότητάς μας να συναλλασσόμεθα μακροπρόθεσμα, να έχουμε βιώσιμο εμπόριο με την Κίνα. Έχετε μια ιδεολογική προσέγγιση κομισιόν. Θα ήθελα να μου πείτε, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, γιατί δεν ήσασταν σε θέση να μας δώσετε, να δώσετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα αμυντικά εργαλεία που έχουν οι Αμερικάνοι για να προστατευθούν. Κύριος Μαρτέο. Νομίζω ότι το θέμα είναι σοβαρό. Οπότε την απόφαση δεν θα πρέπει να την πάρει η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Θα πρέπει να ακουστεί και η φωνή των πολιτών. Και όταν λέω Μιλώ για τους πολίτες, μιλώ για τους πολίτες στο σύνολό τους. Οι εταιρείε, οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι, οι κατανοητές, όλοι θα πρέπει και εμείς να διαβουλευτούμε με έναν τρόπο πολύ πιο ευρύ ε, από αυτόν που ανακοινώσατε εσείς. Ε, πρέπει να είναι κανείς ναΐφ για να ε, αναρωτιέται αν γίνεται dumping, αν υπάρχει ε, το φαινόμενο ε, των επιδοτήσεων, που είναι, το παράνομου επιδοτήσεων κλπ. Το θέμα δεν είναι νομικό, ε, δεν με νοιάζει τι πιστεύουν οι νομικοί. Η απόφαση θα είναι πολιτική. Η πραγματική ερώτηση πρέπει να θέσουμε και το Συμβούλιο θα πρέπει να σταματήσουμε την υποκριτική του στάση. Ο Κάμερον χύνει κροκοδίλια δάκρυα για τις επενδύσεις Ηνωμένο Βασίλειο και από την άλλη μεριά ε, μπλοκάρει το, τον εξυγχρονισμό της εμπορικής μας αμυντικής πολιτικής. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η υποκρισία. Οπότε, σε τι βασίζεστε για να πείτε ότι 250.000 θέσεις εργασία μόνο θα χαθούν. Εγώ πιστεύω θα χαθούν πολύ περισσότερες. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνει μια μελέτη αντικτύπου πολύ πιο σοβαρή. Τελειώνοντας, σας παραπέμπω στην έκθεση του, εμπορικού, του μελητηρίου της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα που λαμβάνει υπόψη ε, ο, πολλούς τομείς, ξύλο, κεραμική, χαρτί κλπ. Ε, έχουμε τεράστιες απώλειες σε θέσεις εργασίας θα έχουμε. Ε, αν οι εξαγωγές της Κίνας έχουν διπλασιαστεί ε, σε 12 μήνες, καταλαβαίνετε γιατί όλοι οι παραγωγοί στην Ευρώπη έχουν ε, ζημιές. Ευχαριστώ, κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως και συνάδελφοι. Και εγώ είμαι κατάπληκτη που θα υποφεληθεί η Κίνα από το ενδιάμεσο αυτό καθεστώ. Επί 15 χρόνια προσπαθούμε να σεβαστούμε κάποια κριτήρια. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα κριτήρια τα σεβάστηκε. Ε, το κοινωνικό κράτο ε, επιδοτεί χοντρά την οικονομία και στον τομέα του χάλιβα, αλλά και σε άλλου. Τα είπαν οι συνάδελφοι. Εάν σήμερα θα έπρεπε να χορηγήσουμε το καθεστώ οικονομική αγορα στην Κίνα, θα χάναμε την ικανότητα που έχουμε να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας. Γιατί οι κανόνε θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να εφαρμοστούν εν τη αυτή περιπτώση. Και οι κυρώσει που θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε θα ήταν πολύ λιγότερο σημαντικές. Επομένως, ούτως ή άλλως όλα αυτά θα κατέστρεβαν ακόμα περισσότερο την ευρωπαϊκή οικονομία που ούτως ή άλλως είναι σε ύφεση και ευθύνη. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν τι τρέχει. Έχετε πάθει τύφλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λειτουργείτε ξανά και ξανά όπως τις προηγούμενες δεκαετίες. Χωρίς να καταλαβαίνετε τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, χωρίς να καταλαβαίνετε τι σκέφτεται ο κόσμος και αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι να υπερασπίσουμε την οικονομία μας. Συγγνώμη, και την βιομηχανία μας θα πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας. Δεν νομίζω ότι υπερασπιζόμαστε τη βιομηχανία μας χορηγώντας στην Κίνα σήμερα το καθεστώ της οικονομίας της αγοράς. Έχω συζητήσει με Κινέζους υπεύθυνου και αξιωματούχου. και του είπα πρέπει να υπάρχει κοινωνική ανάπτυξη στην Κίνα ούτω ώστε κάποια μέρα να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε μια κάποια ισορροπία μεταξύ της Ευρώπης και της Κίνας. Αλλά προς το παρόν είναι αδιανόητο κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται σήμερα να δοθεί το καθεστώς αυτό στην Κίνα. Ίσως σε 10 χρόνια, σε 15 χρόνια, αλλά προς το παρόν είναι αδιανόητο. Θα μας πούνε, ναι θα υπάρξουν αντίπεινα από τους ε, Κινέζους, δεν θα ξαναπολύσετε αεροπλάνα και τα λοιπά στην Κίνα. Πρέπει εμείς να προβλέψουμε τι θα συμβεί. Πρέπει να προβλέψουμε τις συνέπειες, να εφοδιαστούμε με τα κατάλληλα εργαλεία για να υπρασπιστούμε τη βιομηχανία μας, ούτω ώστε να μην υποστεί τις συνέπειες μια τέτοια επιλογή. Η αφέλεια που σας διακατέχει σήμερα είναι τέτοια, λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούμε. Ευχαριστώ κύριε Μπούζεκ. Είπατε γλαφυρά ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε κρίση ακόμα με 40.000 θέσεις εργασίας ε, που διατρέχουν κίνδυνο και ολόκληρες κοινότητες κινδυνεύουν. Ε, μιλήσατε για χάλιβα, γυαλί, κεραμικά. Στο Σεν Τάλλον ήμουν σε μια εκδήλωση στην εκλογική μου περιφέρεια, σε μια μονάδα που διατρέχει κίνδυνο. Μιλήσατε για 250.000 ε, θέσεις εργασίας που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Οι συζητήσεις μας με τα συνδικάτα μιλάνε για νούμερα πολύ μεγαλύτερα, ένα εκατομμύριο. Εμπόριο και βιομηχανία και τα δύο. Χρειάζεται λοιπόν κοινή βιομηχανική στρατηγική για να προστατεύσει τις ε, βιομηχανίες μας που είναι εντατικέ από άποψη χρήσης ενέργειας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε 15 χρόνια. Χρειάζεται ανάληψη δράσης για να σταματήσουν τα προβλήματα τώρα. Ευχαριστώ, συνάδελφο Ταμπουράνο. Θα είμαι λακωνικότατος. με απόλυτα από τις θέσεις που είναι πολύ επικριτικές των προλαλισσάντων. Θα ήθελα μόνο να προσθέσω ότι κατά την άποψη της ομάδας μου θα ήταν σημαντικό το θέμα να συζητηθεί στην Ολομέλεια και να γίνει συζήτηση με ψήφισμα μέχρι το τέλος του μήνα, μια και πιέζουν οι προθεσμίες, ούτως ώστε το Κοινοβούλιο, που είναι το μόνο εκλεγμένο όργανο από τους πολίτες, να έχει τη δυνατότητα να θέσει τη θέση του, να την πει με ξεκάθαρο και μονοσήμαντο τρόπο. Ο πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς. Μια ερώτηση. Ακούσατε όλους τους αδέλφους. Όλοι συμφωνούμε, επικρίνουμε. Ε, επί της ουσίας όμως. Γιατί η Κομισιόν δεν παίρνει ποτέ υπόψη να το Κοινοβούλιο ακόμα και όταν εκφράζεται ομόφωνα. Μία φορά ακόμα δεν θα μας λάβετε υπόψη. Το πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Οικοδόμηση είναι η Κομισιόν. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω και μια δική μου ερώτηση, μια και ολοκληρώθηκε, εξαντλήθηκε ο κατάλογος των ομιλητών. Το πάνελ του ΠΟΕ στις 29 Μαρτίου ε, αμφισβητεί τα μέτρα αντι-dumping για τις αγωγές βιο-δίζελ από την Αργεντινή. Παρόμοια κατάσταση με την επιλογή 3. Έχουμε κάποια εγγύηση ότι ο ΠΟΕ δεν θα αφισβητήσει οποιασδήποτε πρόσθετες, οποιαδήποτε πρόσθετα μέτρα ληφθούν για την Κίνα. Η κυρία Νίμπλερ ε, έθεσε ένα παρόμοιο ερώτημα για την επιλογή 4. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις μας. Θα μπορούσατε να μας απαντήσετε. Ευχαριστώ. Uh, Θα προσπαθήσω να απαντήσω τις ε, πολύ άριθμες ερωτήσεις, όσο μπορώ. Καταρχάς, κάποιες ε, παρατηρήσεις με εξέπληξαν, αλλά συμφωνώ με την ανάλυση του κύριου Λάγκη, ο οποίος μίλησε για τη σημασία των εργαλείων την dumping μίλησε για την σημασία ενός συστήματος το οποίο θα είναι αρκετά ισχυρό ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το ντάμπινγκ της Κίνας. Και είπε επίσης ότι υπάρχουν δύο προβλήματα. Πρώτον, ε, ο εξονισμός των ε, εργαλείων TDI είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να λάβουν δράση τώρα και μια μεταρρύθμιση του συστήματος ε, σε σχέση με την Κίνα, ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τι ε, πρακτικές dumping της Κίνας. Μπορεί να σας εκπλήξει, αλλά να σας τονίσω ότι συμφωνώ απόλυτα με την ανάλυση αυτή. Θέλουμε να έχουμε ένα ισχυρό σύστημα αντι-dumping και στο μέλλον. Ακούστηκε μια ερώτηση γιατί η Κομισιόν δεν έχει, τα, δεν έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοια εργαλεία όπως ε, ε, είπα. Δουλεύουμε με βάση το ενωσιακό δίκαιο. Και από ό,τι ήξερα, από ό,τι ήξερα μέχρι τώρα δηλαδή, και εσείς νομοθέτησαστε. Η κυρία Νίμπλε με ρώτησε τι θα γίνει με τις πιθανές τροπολογίες. Η Κομισιόν θα πρέπει να αποφασίσει καταρχάς αν θα προτείνει η νομοθεσία ή όχι κάνουμε την μελέτη αντικτύπου. Ορισμένοι αποφάσισαν ήδη ποιε θα είναι οι επιπτώσει, χωρί να έχουν κοιτάξει καν την ίδια τη μελέτη. Έχετε το δικαίωμα, το κάνετε βέβαια. Εμεί πιστεύουμε ότι πρέπει να δούμε καταρχά την κατάσταση και πρέπει να κάνουμε μια πλήρη ανάλυση τη κατάσταση και να λάβουμε και τη γνώμη υπόψη των ευρωπαϊκών ενδιαφερομένων πριν ληφθεί απόφαση. Δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση αν θα ε, προτείνουμε νομοθεσία ή όχι. Εμεί ω Κομισιόν δεν έχουμε λάβει απόφαση. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τη μέθοδο υπολογισμού του dumping, θα πρέπει να αλλάξουμε την νομοθεσία πάντω. Και αν αποφασίσει η Κομισιό να υποβάλει πρόταση, τότε η νομοθεσία για αυτά τα θέματα θα υιοθετηθεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Επομένως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει απόλυτα τα προνόμια του ως συνομοθέτης. Μπορούμε να αντιγράψουμε το αμερικανικό σύστημα ενδιαφέρον. Κάποια στιγμή μιλήσατε, είπατε κάτι κυρία Νίμπλερ για τον προστατευτισμό. Είμαστε πολύ περήφανοι για το δικό μας σύστημα, γιατί είναι πιο ισορροπημένο από το αμερικανικό. Και λαμβάνει 100% υπόψη ότι η βιομηχανική πραγματικότητα στην Ευρώπη δεν είναι απλώς η παραγωγή κάποιων προϊόντων. Είναι και οι βιομήχανοι που χρησιμοποιούν τα προϊόντα αυτά και είναι και οι καταναλωτές οι οποίοι καταναλώνουν τα προϊόντα. Και επομένω στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα πολύ πιο περίπλοκο σύστημα που εξετάζει, λαμβάνει υπόψη και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα πριν επιβάλλει μέτρα anti-dumping και τι ζημιά ε, επιβάλλεται και θα πρέπει να διορθωθεί. Το να αντιγράψουμε λοιπόν το αμερικανικό σύστημα φυσικά είναι μια δυνατότητα, αλλά θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι ιστορικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε αναπτύχθηκαν διαφορετικά και οι Αμερικανοί ε, είναι αντικείμενο κριτικής σε μεγάλο βαθμό στον ΠΟΕ. Κύριε Κέρτεν Ντάρλινγκ, ε, τι διάλογο έχουμε. Είμαστε σε επαφή με τους μεγάλους χρήστες ε, του αντι-dumping, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία, Βραζιλία, συγκρίνουμε τις μεθόδους μας, ε, συναντιόμαστε πάρα πολύ τακτικά. Θα γίνει στον ΠΟΕ στο τέλος του μήνα μια επιτροπή αντι-dumping που θα είναι μια καλή ευκαιρία για να συγκρίνουμε τις μεθόδους μας. Και σας λέω από τώρα ότι έχουμε επαφές και σε υψηλότερο πολιτικό επίπεδο με τις ΗΠΑ για το θέμα αυτό. Κάτι που θέλω να τονίσω ξανά είναι ότι σήμερα δεν είμαστε στην ίδια θέση νομικός, νομοθετικός πώς όπως είναι οι Αμερικάνοι. Το θέμα είναι, θα πρέπει να αλλάξουμε το σύστημά μας, ούτως ώστε να ευθυγραμμίσουμε το σύστημά μας με των Αμερικανών. Και αν οι Αμερικανοί αποφασίσουν να αλλάξουν το άλλο το σύστημα. Ξέρετε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν διάφορα θέματα πολιτικού προσανατολισμού που δεν θα ξεκαθαρίσουν πριν αναλάβει η νέα κυβέρνηση του χρόνου, βασικά θα ξεκαθαρίσουν. Υπάρχουν κάποιοι αντικειμενικοί, δηλαδή περιορισμοί, ως προς το, πόσο μπορούμε να συντονιστούμε τους Αμερικανούς. Αλλά είμαστε πάντα σε στενή επαφή με αυτούς. Κύριε Ρίξον, είπε ότι η Κίνα δεν είναι η οικονομία της αγοράς. Το είπα και στην εισαγωγή μου, και εγώ. Είπα όμως ότι δεν πρέπει να γίνει μια συζήτηση για το κατά πόσον η Κίνα είναι τέτοια οικονομία, αλλά αν θα πρέπει να αλλάξουμε τη μεθοδολογία υπολογισμού του ντάμπινγκ. Ο κύριο Έριξον είπε δύο πράγματα, τα οποία είναι πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου. Υπάρχουν δύο προβλήματα. Ε, το πλεονάζον δυναμικό και δεύτερον το dumping. Το πρόβλημα είναι ότι το πλεονάζον δυναμικό τροφοδοτεί το dumping και το υπερβολικό δυναμικό ρίχνει τις τιμές, αλλά και στη χρεοκοπία των επιχειρήσεων. Ε, στην Κίνα δεν υπάρχει νομοθεσία για την χρεοκοπία. Υπάρχει λοιπόν μια σχέση ανάμεσα στο πλεονάζον δυναμικό και στο dumping. Τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το πλεονάζον δυναμικό. Δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσουμε, αλλά το βάζουμε στην ατζέντα σε κάθε συνάντηση που έχουμε με τις κινέζικες αρχές. Έχουμε κάποιες συναντήσεις που γίνονται μέχρι να φτάσουμε στην ε, Σύνοδο Κορυφής. Και γίνεται και μια σημαντική συζήτηση στον ΩΣΑ για το πώς θα αντιμετωπιστεί ε, το πλεονασμαμικό, ή πολλές ε, επιδοτήσεις κτλ. Αλλά το θέμα είναι πολύ πολιτικό σχέση με την Κίνα. Πέρα από τα συστήματα λοιπόν διαλόγου, ε, πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε ε, διάλογο σε υψηλότερο πολιτικό επίπεδο με τους Κινέζους. Κυρία Λόπες Μπερμέχο, μιλήσατε για την απελευθέρωση του εμπορίου. Να μπω σε τεχνικά θέματα εδώ. Όταν μιλάμε για dumping, δεν μιλάμε για την απελευθέρωση του εμπορίου. Δεν μιλάμε για την κατάργηση των δασμών που υπάρχουν σήμερα. Το anti είναι η δυνατότητα να επιβάλλουμε επιπλέον δασμούς. Μπορούμε να επιβάλλουμε επιπλέον δασμούς πέρα από αυτούς που υπάρχουν σήμερα μόνο εάν ε, κάνουμε... Ε, υπάρχει μια διαδικασία. Αν υπάρχει παράπονο, κάνουμε μια έρευνα και συνάγουμε ότι για ένα συγκεκριμένο προϊόν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι, οι νομικοί λόγοι για να επιβάλλουμε επιπλέον δασμούς. Κανένα δεν μιλάει για κατάργηση δασμών που υπάρχουν ούτως ή άλλως απέναντι στην Κίνα. Και αυτό ούτω ε, η άλλω απεναντι στην κινα και αυτο ειναι το μεγαλο λάθο, το μεγαλο προβλημα που εχει αυτη η μελετη ε, που μιλάει για 3,5 εκατομμύρια θέσεων απασχόλησης που μπορεί να χαθούν. Λάθος λέει αυτή η μελέτη ότι μια αλλαγή στη μεθοδολογία του dumping θα μειώσει τους παραδοσιακούς δασμούς που επιβάλλουμε στα κινέζικα προϊόντα συνολικά κα 30% συνολικά. Λάθος είναι αυτό. Απλώς η μελέτη είναι λάθος. Η δική μας μελέτη που την επικρίνατε είναι πολύ πιο σωστή. Γιατί. Γιατί ε, εξετάζει προσεκτικά το τι έχουμε σε δραστηριότητα dumping, δηλαδή τι, δραστηριότητε dumping έχουν, ε, προ, προωθούν οι Κινέζοι. Κύριε Μπορέλη, πώ υπολογίζουμε τι θέσει απασχόληση. Πήγαμε και, εξετάσαμε τα 52 μέτρα που, έχουμε, που τρέχουν κατά τη Κίνα και σε αυτέ τι έρευνε έχουμε λάβει πληροφορίε από την βιομηχανία που παραπονιέται για τι θέσει απασχόληση που σχετίζονται άμεσα με το συγκεκριμένο προϊόν. Σας είπα ότι ο αριθμός των θέσεων απασχόλησης στον τομέα του Χάλιβα είναι 55.000. Εσείς θα μου πείτε αποκλείεται. Γιατί υπάρχουν πολύ περισσότεροι ε, απασχολούμενοι που δουλεύουν στο Χάλιβα στην Ευρώπη. Ναι, σίγουρα. Αλλά αυτοί οι εργαζόμενοι που εντοπίσαμε είναι αυτοί που ε, επηρεάζονται άμεσα από το συγκεκριμένο προϊόν στα πλαίσια της έρευνάς μας. Οι έρευνές μας κοιτάνε πολύ στοχευμένα τον ορισμό ενός ε, προϊόντος. Πάνω σε αυτή τη βάση ε, δουλεύουμε. Για να υπολογίσουμε τις επιπτώσεις. Τι κάνουμε. Κοιτάμε τις παλιές ε, έρευνες, κάνουμε προσωμιώσεις, χρησιμοποιούμε διάφορες μεθόδους. Ε, άκουσα ότι μια αλλαγή της μεθοδολογίας θα καταστρέψει το σύστημα. Έχουμε κάνει και άλλε προσωμιώσει και δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Βλέπουμε ότι με άλλα συστήματα μπορεί να είναι δυνατόν να έχουμε τελικά ένα αρκετά στεναρό σύστημα εδώ στην Ευρώπη. Ε, η δημόσια διαβούλευση ε, είναι πολύ τεχνική. Σωστό. Αλλά το θέμα είναι τεχνικό. Κυρίω αφορά εκείνου που χρησιμοποιούν το αντι και είναι εταιρείε αυτέ που γνωρίζουν πολύ καλά τι είναι και χρησιμοποιούμε Ερωτήσει το κάνουμε και για τι δημόσιε διαβουλεύσει τη εσωτερική αγορά, γενικά. Εγώ δούλεψα, δούλευα στις επενδύσεις και είχα κάνει μία δημόσια διαβούλευση ε, για τις επενδύσεις με ανοιχτές ερωτήσεις, όχι κλειστές ερωτήσεις. Και όμως με επικρίνανε και γι' αυτό, ότι με αυτόν τον τρόπο η Κομισιόν λέει ε, δεν είναι μερόληπτη. Ε, τι να σας το πω. Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Προσπαθούμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το Πανεπιστήμιο της Λουβέν πήρε τη μελέτη και οι όροι του συμβολέου ε, έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης ε, Εμπορίου. Το Πανεπιστήμιο του Λουβέν είναι από τα καλύτερα και τα παλιότερα της Ευρώπης. Και αυτό έχει κάνει λοιπόν τη μελέτη, ήθελα να το πω. Νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Η τελευταία ερώτηση του Πρόεδρου για το βιοντίζελ της Αργεντίνα, Αργεντινής. Ε, είναι λίγο διαφορετικό το θέμα. Εδώ θα πρέπει να αποφασίσουμε εάν θα έχουμε λόγο να προσαρμόσουμε ένα στοιχείο του κόστους. Δεν είμαστε πεπισμένοι από την επιχειρηματολογία του πάνελ του ΠΟΕ. Εδώ μιλάμε για μια πολύ γενικότερη συζήτηση, ένα πολύ γενικότερο θέμα μεθοδολογικό. Υπάρχουν ομοιότητες, αλλά θα χρησιμοποιήσω αυτό το πάνελ για να, για να συνάγω τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον ε, για την Κίνα. Μακρηγόρησα, αλλά και οι ερωτήσεις ήταν πάρα πολλές. Εμείς τις χρειαζόμαστε όλες τις ε, απαντήσεις γιατί είναι σημαντικές οι ερωτήσεις και είναι σημαντικό το όλο θέμα της χορήγησης του καθεστώτος οικονομίας αγοράς στην Κίνα. Πολύ σημαντικό για την οικονομία μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Διευθυντά. Σας ευχόμεθα κάθε επιτυχία και να ακούτε και τη δική μας τη φωνή. Αυτό είναι σημαντικό για όλους μας. Ευχαριστώ και πάλι. Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, τώρα προχωρούμε στο σημείο 5, δηλαδή ψηφίζουμε. Καταρχήν να κάνουμε μια δοκιμή. Ψηφίζουμε δοκιμαστικά. Πάρτε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες παρακαλώ. Uh, λοιπόν, τοποθετήστε συσχισμή σχισμή την κάρτα. Είναι σημαντικό αυτό που κάνουμε. Now uh, is a Λοιπόν, ψηφίζουμε δοκιμαστικά. Τι ερώτηση να βάλουμε. Ε, ε, αγοράσατε το εισιτήριο επιστροφής σας. Αυτό είναι που θα ψηφίσουμε. Με ναι ή όχι. Έτσι. Ψηφίζουμε δοκιμαστικά. Και νομίζω ότι είναι και πολύ ε, καλό το ερώτημα. Ενδιαφέρον. Πέρα της ψηφοφορίας. Θαυμάσια. Όμως πρέπει να παραμείνετε μέχρι τις 6.30 σήμερα το απόγευμα, γιατί τότε λίγη η συνεδρίασή μας. Εντάξει, τώρα θα πάμε στην καθαυτό ψηφοφορία. Ανταγωνιστικότητα του Ευρωπαϊκού Κλάδου Προμήθεια ιδροδρομικού Υλικού, Μαρτίνα Βέρνερ, είναι η συγκήτρια. Προφορική ερώτηση, έχουμε μία μόνο ψηφοφορία να κάνουμε εδώ. Ε, ηλεκτρονικά όμως θα ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. δεκτή. Uh, well, okay, okay. Oh, okay. Εντάξει, επαναλαμβάνουμε, αγαπητοί φίλοι. Εντάξει γιατί έχει δυσκολίες, έχουν δυσκολίες οι Βρυξέλλες σε αυτή την εποχή. Αρχίζει η ε, ψηφοφορία, αυτό που ψηφίσαμε, ανταγωνιστικότητα του Ευρωπαϊκού Κλάδου, το σημείο 5. Λοιπόν, όλοι εντάξει ψηφίσατε, πέρας. Πολύ καλύτερο το αποτέλεσμα τώρα. Δεκτή. Και προχωρούμε τώρα. Πρόταση ψηφίσματος κυρία Μαρτίνα Βέρνερ, πάλι για την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου. Τροπολογία 14, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές ε, ηλεκτρονικός έλεγχος 31 έναρξη ψηφοφορίας Λήξη ψηφοφορίας. Γίνεται δεκτή. Παρακαλώ σηκώνετε το χέρι σας. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται, αλλά ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Η 48. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 53. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος ή 60 τροπολογία 60 λίγη ψηφοφορία απορρίφθηκε 62 υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος. Για την 62. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 70 και 80 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 75 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για την 75 Open the vote. Λίγη Εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 107 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 12 υπέρ όχι ε, ηλεκτρονικός έλεγχος της 107 ηλεκτρονική βεβαίωση για την 107 έρχεται η ψηφοφορία λήξη ψηφοφορίας απορρίπτεται Παρακαλώ σηκώνετε το χέρι σας για να σα βλέπω. Ε, αυτό είναι το δικό μου, ο δικό μου καημό. Συμβαστική 12, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 117 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16 με την τροπολογία των πρασίνων. Τη γνωρίζετε, είναι προφορική τροπολογία. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια αντίρρηση. Υπάρχει αντίρρηση να ψηφιστεί. Εφόσον υπάρχει αντίρρηση, δεν ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία των πρασινών. Συμβαστική πρόταση 16 χωρίς την προφορική τροπολογία των πρασινών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 137 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επιβεβαίωση. 137. Λήξη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβασμό συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 146. Όχι. Ε, έχουμε προφορική τροπολογία από το ΕΛΚ. Έχετε αντιρρήσει. Ναι, ναι. Βλέπω αντιρρήσεις. Οπότε ψηφίζουμε την 146 χωρίς την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 153 λέει ο πρόεδρος. Υπέρ. Η 152 έγινε δεκτή. Οπότε θα πρέπει να περάσουμε στην 153. Οπότε σας, ζητώ, σας ρωτώ για την 153. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. ηλεκτρονική επαλήθευση. Για την 153. Λήξη της ψηφοφορία εγκρίνεται. Συμβασμός 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 156. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 165. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 167. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 169 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 170 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 174 υπέρ. Κατά. ηλεκτρονική επαλήθευση. Για την 174. λήξη της πληροφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 178 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 180 υπέρ. Α, δεύτερο τμήμα. Μόνο το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 182 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 190 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 191 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 192 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 23, συμβασμός 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 210 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 211 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 212 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβασμός 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 218 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 218 λήξη της πληροφορίας εγκρίνεται συμβασμός 26 20, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 224 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 222 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 226 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 227 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται νομίζω τουλάχιστον θέλετε ηλεκτρονική επιβεβαίωση η ηλεκτρονική επιβεβαίωση για τη 227 λήξη της πληροφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για την 13 λήξη εγκρίνεται τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά έναρξη της ψηφοφορίας για το σύνολο του ψηφίσματος. Λήξη της φοφορίας. 51 ψήφοι υπέρ, 6 κατά. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια στην κυρία Μπέρνερ. Περνάμε στο δεύτερο κείμενο. Μια νέα μακρόπνονη και καινοτόμως μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις της κυρίας Γκρίφιν. Έκθεση κυρίας Γκρίφιν εκ μέρους της Επιτροπής Ήτρε. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 14 λήξη ψηφοφορίας απορρίπτεται με 16 εποχές. 15 υπέρ. Κατά. εποχές Απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. εποχές Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. εποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 5 ποιος είναι υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση συμβαστική 5 λήξη Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Για την 46. Συγγνώμη. Για την 34. Για την 34. Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για 49 λήξεις ψηφοφορίας απορρίπτεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Για την συμβαστική 9. λήξη τη ψηφοφορίας εγκρίνεται. 63. Τροπολογία 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75. Εδώ έχουμε προφορική τροπολογία από τους σοσιαλιστές ε, και τους δημοκράτες. Υπάρχει αντίρρηση? Ναι. Υπάρχουν αντιρρήσει, άρα η ψηφοφορία γίνεται χωρί την προφορική τροπολογία. Τροπολογία 75 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 77 υπέρ. Ε, όχι. Ε, επαλήθευση για την 75. Πολύ καλά. Επαλήθευση για την 75. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για την 77 λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά Αποχές. Επαλήθευση για την 79. Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση για την 82. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. 84. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Λήξη τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 86. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Επαλήθευση. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 86. Λήξη τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 87. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση για την 87. Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο του ψηφίσματος. Λήξη ψηφοφορίας. 48 υπέρ 6 κατά 3 αποχές. Συγχαρητήρια. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Ε, Μάριαν Ζαν Μαρινέσκου. Διαστημικές δυνατότητες συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 9, προφορική τροπολογία από την εισηγήτρια και την κυρία Κρέλ. Έχετε αντίρρηση? Δεν έχει κανείς αντίρρηση. Ωραία. Η 9 λοιπόν, μαζί με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή, 13 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 14 υπέρ. Α, έλεγχο στη 13, ωραία, ψηφίζουμε τη 13 ηλεκτρονικά. Πέρας. Δεκτή η 13. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 15. Υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 33 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 44 υπέρ το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 56 υπέρ κατά αποχές έλεγχος, έλεγχος στην 56 Ψηφίζουμε την 56 τροπολογία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 62 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Αγαπητοί σοσιαλιστές συνάδελφοι, σηκώνετε το χέρι, πλησιάζουμε στο τέλος. 62, ψηφίζουμε την 62. Έλεγχος ηλεκτρονικός θα γίνει. Πέρας. Απερίφθη. Τώρα, ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία ε, τελική. Πέρας. Το αποτέλεσμα είναι θετικό. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Διαστημικές δυνατότητες για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα. Αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν το σημείο 5, 6 και 7 στην ημερήσια διάταξη. 5, 6 και 7 είχαμε. Και τώρα πάμε στο σημείο 8, στην ώρα μας ακριβώς, ακριβώς στην ώρα μας, 10 και 30 είναι η ώρα. το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, προβληματισμοί για το πρώτο έτος λειτουργίας και τη μελλοντική πορεία, ανταλλαγή απόψεων με το Διευθύνοντα Σύμβουλο Βίλχελμ Μόλτερερ. Αγαπητοί φίλοι, είμαστε ακριβώς στην ώρα μας, αλλά δώστε μας τη δυνατότητα να αρχίσουμε. Δεν θέλετε να παραμείνετε Ωραία. Αφού δεν θέλετε, μία δυνατότητα είπα, έχετε ή να μείνετε ή να είστε ήσυχοι. Δεν με ακούει κανείς όμως. Well, I Όπως το δημοτικό. Θα κάνω το δάσκαλο της πρώτης δημοτικού. Λοιπόν, το θέμα μας. Να σας το επαναλάβω. Οι συνάδελφοι Τούρμες και Βαν Μπρέντ, παρακαλώ. Δεν, δεν Δεν μ' ακούνε καθόλου. Συνάδελφε Λάνε, συνάδελφε Ρόιλ, συνάδελφε Λάνεν. Παρακαλώ, πείτε τους κάποιος. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα μας είναι πολύ σημαντικό. Το έτσι. Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, προβληματισμοί για το πρώτο έτος λειτουργίας και τη μελλοντική πορεία. Ανταλλαγή απόψεων με το Διευθύνοντα Σύμβουλο Βίλχελμ Μόλτερερ. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κανονισμός ε, εδώ εγκρίθηκε το 2015 και εμείς ασχοληθήκαμε πολύ διότι ισχύει ο κανόνας 54 και δίνει αποκλειστικές αρμοδιότητες. Ο εισηγητής μας δεν είναι μαζί μας. Πάντως επρόκειτο για την πηγή χρηματοδότης και την πλειοψηφία των τομέων επενδύσεων. Το Ταμείο και η δομή του τώρα έχουν συσταθεί και με ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγης την εφαρμογή, την πρακτική υλοποίηση του μέσου. Χρειάζονται χρήματα, όχι πολλά ευτυχώς, γιατί εμείς τα χρήματά μας τα θέλουμε να δοθούν στο Horizon 2020. Όσα είναι να ε, δοθούν πρέπει να δοθούν. Και έχουμε επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια. Όμως, παρόλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι θέλουμε να δούμε τα αποτελέσματα μετά από ένα χρόνο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Αυτού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, του ΕΤΣΕ στα ελληνικά. Λοιπόν, κύριε Διευθυντά, δώστε μας ε, τα καινούργια στοιχεία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, καλημέρα σε όλους, είναι χαρά που είμαι εδώ. Θα κάνω στα γρήγορα μια εισαγωγική παρουσίαση. Καταρχήν να θυμηθούμε ότι στην Ευρώπη ακόμα έχουμε χαμηλή ανάπτυξη και το ποσοστό ανάπτυξης είναι λίγο. Έχουμε μια κατάσταση στην απασχόληση που είναι ε, μη ικανοποιητική, ιδιαίτερα δυσάρεστη, ιδιαίτερα αν δούμε κάποιες περιφερειακές χώρες και αν δούμε και τους νέους. Τρίτον, υπάρχει κοινό επενδυτικό στην Ευρώπη ακόμη, παρόλο που έχουμε κάποια βελτίωση, ακόμα υπολοιπόμεθα κατά πολύ του επίπεδου του 2008, πριν από την κρίση δηλαδή, και τέταρτον, για την μακροπρόθεσμη προοπτική είναι κλειδί αυτό, έχασε ανταγωνιστικότητα η Ευρώπη σε σχέση με τους διεθνείς ανταγωνιστές. Τώρα, ποια είναι η εμπειρία αγοράς μας σε αυτή την κατάσταση, Πρώτα απ' όλα οι πελάτες, οι επιχειρηματίες παραπονιούνται για την ε, κανονιστική αβεβαιότητα στην αγορά και η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια ε, είναι πρόσκομα για τις επενδύσεις. Δεύτερον, έχουμε ε, περιορισμένη δυνατότητα ανάληψης κινδύνου από τις εμπορικές τράπεζες ε, εν για, ε, ε, αυτό ισχύει από πριν από την Τραπεζική Ένωση. Επίσης είναι δύσκολο να δοθούν δημόσιες, να γίνουν δημόσιες επενδύσεις και δαπάνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ακόμα ε, αναπτυγμένη κέφαλη αγορά σε σχέση με άλλους ανταγωνιστές και παράλληλα έχουμε και υψηλή ρευστότητα στην αγορά υψηλότερη από αλλού και με βάση τις δραστηριότητες της ΕΚΤ. Γι' αυτό αυτό το επενδυτικό σχέδιο το άρχισε ο πρόεδρος Γιούγκερ και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να σας θυμίσω ότι αυτό το επενδυτικό σχέδιο στηρίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι η δημιουργία περιβάλλοντος φιλικού στις επενδύσεις, να βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα, να ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά, η ψηφιακή αγορά, η ενεργειακή αγορά, η Ένωση Κεφαλαιαγορών για να, και να γίνουν διαθροτικές αλλαγές στα κράτη-μέλη και να απομακρυνθούν τα εμπόδια. Δεύτερος πυλώνας, υποστήριξη των επενδύσεων και της πραγματικής οικονομίας ε, και επενδυτικά ε, και συμβουλευτικά. Ε, ήδη αυτό γίνεται από τον περασμένο Σεπτέμβρη, είναι κέριο θέμα και επίσης υπάρχει και μία πύλη που ε, φροντίζει για την σωστή ενημέρωση και προετοιμασία. Τρίτος πυλώνας, κινητοποίηση ε, μέσων χρηματοδοτικών και πρόσβαση σε αυτά για την πραγματική οικονομία. Αυτό είναι το περίφημο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων που είμαι ο Διευθύνων Σύμβουλος και αυτό έγινε και με απόφαση δική σας. Πού βρισκόμαστε τώρα. Καταρχήν, η διακυβέρνηση του Ταμείου από την 1η Ιανουαρίου φέτος έχει, λειτουργεί πλήρως. Δεν έχουμε μόνο δηλαδή το ε, Συμβούλιο, έχουμε και την ε, Παιδιτική Επιτροπή και έχουμε και το Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα άλλα μέλη έχουν αναλάβει πλήρως καθήκοντα. Έχουμε σαφή καθοδήγηση για τη δραστηριότητά μας. Έχουμε καταρχήν δηλαδή τον κανονισμό που εγκρίθηκε από εδώ και το είπατε ότι ήταν μια πάρα πολύ ταχεία διαδικασία. Ο κανονισμός δίνει σαφείς ενδείξεις και προσανατολισμούς για το τι είναι επιλέξιμο, την προσθετικότητα, όλα αυτά τα σχετικά τα λέει. Γι αυτό, αυτό είναι το κλειδί για μας. Επίσης, εντωμεταξύ πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι πρόσθετοι κανόνες που θεσπίστηκαν από το Εκτελεστικό Συμβούλιο που διέπει τη δραστηριότητά μας ε, και τη δουλειά μας στην Επενδυτική Επιτροπή. Υπάρχει στρατηγικός προσανατολισμός, υπάρχει ο λειτουργικός προσανατολισμός για το Ταμείο, επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές, η μεθοδολογία, τους βασικούς δείκτες απόδοσης και τη μεθοδολογία ε, που στηρίζεται σε αυτούς. Είναι ένα έγγραφο πολιτικής ε, που υπάρχει για συνεργασία με επενδυτικές πλατφόρμες και επενδυτικές τράπεζες και επίσης ε, αυτό μας καθοδηγεί σχετικά με τις επενδύσεις ταμεία των ταμείων. Είναι σημαντικό να ξέρετε ότι όλα αυτά τα έγγραφα είναι δημόσια, είναι ανοιχτά και προσβάσιμα. Και η τρίτη κατευθυντήρια γραμμή είναι ο πίνακα επιδόσεω, όπου εδώ το Κοινοβούλιο έκανε μεγάλη προσπάθεια για να αναβαθμίσει την ποιότητα του πίνακα επιδόσεων, αυτό για την αξιολόγηση το, του τέταρτου πυλώνα, του, και αυτό είναι πολύ βασικό. Ε, τέσσερις πυλώνες λοιπόν, συμβολή στους στόχους του έτσε, τους ξέρετε, στηρίζονται και στον κανονισμό. Δεύτερος πυλώνας είναι η ποιότητα του έργου. Τρίτον, τεχνικά θέματα και ε, οικονομικά. Και το τέταρτο είναι ο πίνακας επιδόσεων, οι δείκτες... Ε, που αφορούν ε, την προσθετικότητα, ε, τη συγκέντρωση χρημάτων ε, από πολλές πηγές. Έτσι λοιπόν δουλεύουμε. Πού βρισκόμαστε τώρα μετά το εννιάμινο εφαρμογής του έτσε. Εν τω μεταξύ αποφασίσαμε Ε, σχετικά με 10,5 δις χρηματοδότηση επενδύσεων που στηρίζονται από το έτσι. Ε, δίνουμε κίνητρα ε, σε 78 δις ευρώ έτσι. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε στο 25% του στόχου που είχαμε των 315. Καλύπτουμε μέχρι το τέλος Μαρτίου 24 από τα 28 κράτη-μέλη. Ε, αυτό με βάση την Τράπεζα Επενδύσεων ε, έχουμε την, και, και, τις καινοτομίες και το, τις μικρομεσαίες που καλύπτονται από το Ταμείο ε, Επενδύσεων. Οπότε σε συνδυασμό γίνεται καλά η δουλειά. Αυτό που είναι επίσης σημαντικό είναι ότι στο, στην κατανομή των τομέων ε, έχουμε κάποιες προτεραιότητες όπου η μία σίγουρα είναι η ενέργεια, η ενεργειακή απόδοση, και ενεργειακή κατανομή. Ε, δεύτερο τομέα οι μεταφορές, όλες οι επενδύσεις στην ε, υποδομή των μεταφορών. Τρίτο, τρίτη προτεραιότητα είναι η υποστήριξη των ΜΜΕ στην Ευρώπη, το περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και καινοτομία και θα υπάρχει και θα, θα σας δοθεί και μια διαφάνεια όπου βλέπετε ένα μικρό κομμάτι. Αυτό είναι ε, για έρευνα και ανάπτυξη. Υπάρχει έρευνα και ανάπτυξη παντού. Ε, υπάρχει σε όλους τους τομείς ε, έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομίες. αυτό που θα δείτε λοιπόν ως έκθεση αργότερα στη διάρκεια του χρόνου θα σας δώσει μια πολύ σαφέστερη και εστιασμένη εικόνα και θα δείτε ότι οι στόχοι αύξησης της ικανότητας και στην έρευνα και στην ανάπτυξη και στην καινοτομία δεν είναι ε, μόνο λόγια, είναι και πρακτικές ε, ε, αποτελεσματικές. Πρέπει να μιλήσω και για τη μελλοντική πορεία, ποιες είναι οι προκλήσεις. Θα παρουσιάσω έξι σημεία και για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει τώρα. Καταρχήν δημιουργία έργων. Εμείς δεν είμαστε ο θεσμός που φτιάχνει τα ε, προγράμματα, εμείς τα, τα ε, ε, χρηματοδοτούμε με βάση τη, αυτό που θέλει η Τράπεζα Επενδύσεων. Χρειάζονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, εδώ είναι και η πύλη που έχει δημιουργηθεί ε, σαφής στόχο για τον επόμενο μήνα να καλύψουμε και τα 28 κράτη-μέλη. Είναι σαφής ο στόχο. Πρέπει να είμαστε ε, ενεργοί, να έχουμε παρουσία σε όλα τα κράτη-μέλη. Τρίτον, θα πρέπει να αυξήσουμε τη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών. Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό το θέμα. Θυμάστε στην αρχή του εγχειρήματο τις συζητήσει που έγιναν για την τον περίφημο κατάλογο των έργων. Ε, δημιουργήθηκε η εντύπωση τότε ότι το εγχείρημα αφορά τις δημόσιες υποδομές. Όχι. Το εγχείρημα είναι να εξισορροπήσουμε ε, ιδιωτικές επενδύσεις και δημόσιες επενδύσεις. Θέλουμε από τις να καλύψουμε νεοφυείς και μεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να ε, καλύψουμε το, τις εγγύησεις ως ταμείο και για τη χρηματοδότηση των υποδομών πρέπει να καλύψουμε το κενό που υπάρχει σε επίπεδο κρατών μελών για τη δομημένη χρηματοδότηση και να έχουμε και για τις δημόσιες υποδομές ε, συγκέντρωση κεφαλαίων από πολλές πηγές και μια κοινή πρόκληση είναι να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τη δυνατότητα ανάμειξης ε, που υπάρχουν μεταξύ δραστηριότητας ε, έτσι και τα διαρθρωτικά ταμεία. Εδώ υπάρχει μεγάλη δυνατότητα να συνδέσουμε τα διαφορετικά ταμεία, ταμεία συνοχής, δεύτερο πυλώνα, με το έτσι για να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα αυτή τη δυνατότητα ανάμειξη που υπάρχει και τη σχετική φιλοσοφία. Όχι μόνο με τα συγκεντρωτικά κονδύλια, αλλά και τα αποκεντρωμένα κονδύλια από τα διαφορετικά ταμεία. Τελειώνω εδώ και θα είμαι ευτυχής να απαντήσω στις ερωτήσεις σας, αλλά όχι μόνο για σήμερα. Αν σας ενδιαφέρει να συνεχίσουμε τις συζητήσεις και τις επικοινωνίες, θα είμαι ευτυχής να ανταποκριθώ σε μελλοντικέ σας προσκλήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τα εισαγωγικά σας λόγια. Τις πολιτικές ομάδες τώρα, από το ΕΛΚ καταρχήν. Ο κύριος Κάριντς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ για την σύντομη και εύληπτη παρουσίασή σας και την περίληψη που μας δώσατε, πολύ χρήσιμη. Έχω μια-δυο ερωτήσεις που πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Πρώτον, δηλαδή, τα ποσοστά στις, ε, στην ενέργεια, στις μεταφορές κτλ. Τα, τα ποσά που πηγαίνουν είναι περίπου τα ίδια, αυτό που έχει συμφωνηθεί. Πότε προβλέπετε θα φτάσετε το 100% της χρηματοδότησης. Πού ήταν ο στόχος ε, που είχαμε συμφωνήσει όταν ε, δημιουργήσαμε το ΕΦΣΥ. Τρίτον, υπάρχει σταθερό ενδιαφέρον, αυξάνεται, μειώνεται. οι ιδιωτικοί επενδυτές ε, δείχνουν ενδιαφέρον ε, με βάση τα κριτήρια που έχουμε θέσει. Εγώ θα πρέπει να πάω στην διάσκεψη των Προέδρων σε λίγο, στις ακριβώς. Θα φύγω λοιπόν ε, από τη συνεδρίαση. Δεν υπάρχει κανένας αντιπρόεδρος παρόν, αλλά έχουμε τον παλαιότερο ευρωβουλευτή, όχι τον γυρεότερο, τον παλαιότερο, που είναι ο κύριος Ρούμπικ και τονίζω όχι ο γυρεότερος. Θέλω να ε, προεδρεύσει στη συνεδρίασή μας μέχρι τις 1.30. Η Αμούντι θα πάρει το λόγο. Ε, εκπροσωπώ και την Κάθριν Λαμπρέντ που δεν μπορεί να έρθει εδώ. Βαν Μπρέντ, Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Με χαρά σας βλέπω εδώ και χαίρομαι που προσφέρεστε να επανέλθετε στη συνεδρίασή μας, στην ε, Επιτροπή μας. Θα ξέρετε ότι αυτή η Επιτροπή είναι υπεύθυνη που βοήθησε να θεσπιστούν οι προτεραιότητες του ΕΦΣΥ και το πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτό το ταμείο. Ε, είναι πολύ χρήσιμα αυτά τα κονδύλια, πολύτιμα αυτά τα κονδύλια ε, που σειραίων προς το ΕΦΣΥ θα προσπαθήσουμε να τα διατηρήσουμε. Από τις προτεραιότητες που θέσαμε υπήρχε η καινοτομία, αναφερθήκατε σε αυτήν, την απόλυτη καινοτομία, την υψηλή προστιθέμενη αξία, δηλαδή υψηλή προστιθέμενη αξία των έργων, βοήθεια των επίτευξη των στόχων εν έρευνας, κλίματος, καταπολέμησης κλιματικής αλλαγής, δεδομένης και της Συμφωνίας του Δεκεμβρίου. Με βάση τα όσα έχουμε πετύχει τώρα στην, στην αρχική φάση. Δεν είμαστε σίγουροι κατά πόσο οι στόχοι που έχει θέσει η Επιτροπή μας έχουν υλοποιηθεί, ειδικά στην καινοτομία και στην βιωσιμότητα. Καταλαβαίνω τι λέτε εσείς, αλλά με ανησυχεί λιγάκι ότι ο ορισμός του, της καινοτομίας έχει έτσι λίγο χαλαρώσει, έχει απλωθεί τόσο πολύ, ε, που δεν ξέρω κατά πόσο, να πούμε, υλοποιούμε το στόχο. Η αξιολόγηση και ο πίνακας επιδόσεων για τον οποίο μιλήσατε θα πρέπει να είναι δημόσιοι δημόσια πράγματα, στο δημόσιο τομέα, να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Θα πρέπει να χρησιμοποιεί το πίνακα αυτό ε, αποτελεσμάτων με πιο α, διαφανή και ανοιχτό τρόπο. Επίσης, πριν η Επενδυτική Επιτροπή δημιουργηθεί, ε, η Κομισιόν έδωσε το OK. Υπάρχουν λίγα προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητα κατά την απόψή σα. Επίση, στο τέλο τη παρουσίασή σα μιλήσατε για το πρόβλημα ορατότητας που έχετε σε ό,τι αφορά απέναντι δηλαδή στους και στους δημόσιους όμως επενδυτές. Και τέλος, για τις πλατφόρμες. Όταν κοιτάμε το ΕΦΣΥ, το πώς θα θεσπιστούν οι πλατφόρμες και το πώς θα αναπτυχθούν ε, και πώς θα συγχωνευτούν διάφορα μικρότερα ενέργεια, ε, έργα ε, με έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά και διάφορα συνεργατικά μοντέλα, πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Γιατί η ενέργεια είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα που η συνεργασία μπορεί να δώσει καλά αποτελέσματα. Ο Κλοντ Τούρμες είναι ο επόμενος. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που έχουμε ένα πεπειραμένο άνδρα που χειρίζεται το ΕΦΣΥ. Ήταν τεράστια οργανωτική πρόκληση να, το να βρούμε τους κατάλληλους ανθρώπους για να το χειριστούν το ταμείο αυτό. Μία ερώτηση που ίσως η Κομισιόν θα πρέπει να απαντήσει περισσότερο. Εμείς, εμάς μας υποσχέθηκαν ότι θα έχουμε 300 εκατομμύρια και πάνω για τεχνική βοήθεια. Μετά την ψηφοφορία μας ανακάλυψα ότι η Κομισιόν δεν μας είχε πει την πλήρη αλήθεια. Στην πραγματικότητα έχουμε 20 εκατομμύρια. Και βλέπουμε το τι λέτε εδώ και τα όσα υπόθηκαν στη συζήτηση. Μιλάμε για βοήθεια, τεχνικής βοήθειας από τα διαφορετικά ταμεία. Τα ταμεία που τα υπολόγισε η Κομισιόν, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα λεφτά δεν θα είναι στις Βρυξέλλες, αλλά ότι έχουν μοιραστεί ήδη. Το πρόβλημα που είχαμε λοιπόν και με την ενεργειακή αποδοτικότητα είναι ότι εσείς είχατε δυόμιση, περίπου τρεις ε, εμπειρογνώμονες για ενεργειακή αποδοτικότητα που θα βοηθούσαν για να ε, ομαδοποιηθούν έτσι τα, τα έργα. Έτσι. Είναι σημαντικό, γιατί έχουμε πάρα πολλά κατακαιρματισμένα έργα και θα πρέπει κάποια στιγμή κάπως να συγχωνευτούν. Αλλά με τρεις εμπειρογνώμονες, ε, αυτό ομολογήσουμε, δεν μπορούμε να ε, δημιουργήσουμε το δυναμικό που χρειάζεται, να το συγκεντρώσουμε. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να φτιάξουμε την απαραίτητη ορμή την απαραίτητη όθηση, ούτω ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα λεφτά από τα διαφορετικά ταμεία για την τεχνική βοήθεια, ούτω ώστε να πληρώσουμε την τεχνική βοήθεια. Εγώ πρότεινα ήδη το Σεπτέμβριο και στην ε, EIB, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στην Κομισιόν, ένα μοντέλο για την Νότια Ευρώπη, να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο ε, για την νότια Νοτιοανατολική Ευρώπη, για την τεχνική αγωγή, με τεχνική πραγματογνωμοσύνη από την ΑΕΠ που θα παίρνουν λεφτά για να πληρώσουν για εμπειρογνώμονες Ρουμάνους, Σλοβαίνους, Βούλγαρους κτλ. Ε, η Νοτιοανατολική Ευρώπη και οι κυβερνήσεις της συμφώνησαν με αυτό το μοντέλο. Κομισιόν, πέστε μου, είναι καλή ιδέα σήμερα αυτή. Ή θα μου πει, ή πέστε το, αν θεωρείτε ότι είναι σαχλαμάρα, ξεκάθαρα. Γιατί δεν μπορώ να λαμβάνω Twitter από τον κύριο Σεύκοβιτ ε, που μου λέει τέλεια ιδέα σα και μετά από έξι μήνε δεν έχει γίνει τίποτα για το θέμα αυτό. Η Ανατολική Ευρώπη. Η Πολωνία ε, έχει ένα μεγάλο κομμάτι από τα λεφτά. Αλλά από πρώτη ματιά είδα ότι είναι αναλογικά λιγότερα τα λεφτά από ό,τι προβλεπόταν. Έχετε ε, απάντηση αυτό και μπορεί η τεχνική βοήθεια να είναι τμήμα τη απάντηση. Ο κύριος Κατάιναν ήρθε και είπε ότι θα υπάρχει ε, μία δικτυακή πύλη για τα έργα. Πού είναι, πού έχετε φτάσει τεχνικά. Ε, την προχωρείτε αυτή την πύλη. Στη διαφάνειά σα λέτε ότι είναι 7,5 η μόχλευση. Ενώ στις συζητήσει πόσο ήταν. 15 και. Είμαστε σκεπτικιστές και εγώ και ο κύριος Δεμπάκ. Σας παρακαλώ, δώστε μας λιγάκι περισσότερα στοιχεία για αυτό το θέμα. Ο κύριος για την προσθετικότητα και την πολλαπλασιαστικότητα θα πρέπει να μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα τι συμβαίνει. Ε, αυτά που είδα, τα project που είδα εγώ, τα έργα που είδα εγώ ήταν αυτά που είχαν, είχε επιλέξει η Ευρωπαϊκή η Τράπεζα Επενδύσεων, ε, πιο παραδοσιακά προγράμματα. Ε, ποια είναι τα νέα έργα τα οποία επιλέχθηκαν που υποτίθεται θα είναι μεγαλύτερου επιχειρηματικού κινδύνου, θα βασίζονται πιο πολύ ε, στην συμμετοχή των ιδιωτών και μετόχων κλπ. Δεύτερη ερώτηση σχετική. Το είπατε κι εσείς ότι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα ενδεχομένως υστερεί λίγο σε σχέση με αυτό που θα περιμέναμε. Πώς θα το διορθώσετε. Γιατί προφανώς στην αρχή τα κράτη-μέλη ζητούσαν 100% κρατική χρηματοδότηση. Πρέπει όμως να έλξουμε περισσότερο, οι περισσότερους ιδιώτες. Ε, μήπως θα πρέπει να το εξετάσουμε περισσότερο, να δούμε πώς θα τους έλξουμε, έστω και καθυστερημένα. Πώς θα τους προσελκύσουμε. Τώρα, για τις διάφορες πλα... επενδυτικές πλατφόρμες, οι οποίες αρχικά κατασκευάστηκαν με στόχο να εμπλακούν ιδιώτες επενδυτές. Κατά την άποψή μου, έτσι όπως το βλέπω εγώ, είναι πιο πολύ κρατικές πλατφόρμες στις οποίες συμμετέχουν σε κάποιο μικρό βαθμό και ιδιώτες. Οπότε, τι γίνεται και εδώ έχουμε τον κρατικό τομέα, το δημόσιο τομέα, ο οποίος είναι μπροστά, μπροστάρις και οι ιδιώτες υστερούν. Μήπως θα πρέπει να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες στους ιδιώτες. Τρίτον, το, τα έργα σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, ο κ. Κατάινεν πάντοτε μας έλεγε ότι η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι σημαντικό κομμάτι. Όμως ε, θέλουμε οι επενδύσεις να είναι μεγαλύτερο κίνδυνο και να βασίζονται σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Όμως βλέπουμε ότι μεγάλα ποσά ε, χρησιμοποιούνται για την ε, ε, επενδυτική ενίσχυση των τραπεζών, αλλά οι τράπεζες από μόνες τους δεν θα βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς θα πρέπει τα χρήματα του Ταμείου να πηγαίνουν κατευθείαν σε κάποιο βαθμό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι ώστε να αφαιρέσουμε λίγο από τα προβλήματα των, των τραπεζών που είναι προβλήματα ε, ε, χρευστότητας. Από την ε, Γκουε τώρα, η κυρία Λόπες Βερμέχο. Έχω την εντύπωση ότι τα ταμεία σας δεν επιτυχάνουν και πολύ, οι, συγγνώμη, οι πόροι σας δεν έχουν μεγάλη επιτυχία στην Ισπανία. Ε, τα κονδύλια αυτά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ στην Ισπανία. Ε, τα ομόλογα έργου ε, έχουν χρηματοδοτήσει το Κάστορ που έχει χάσει χρήματα 1,8 δις μάθαμε τελευταία και τώρα χρηματοδοτείται η Αβενγκόα ε, μέσω της οποίας χάνει η Τράπεζα Επενδύσεων άλλα 4 δις. Οπότε η ερώτηση είναι εξή. Ποιο τμήμα αυτών των απολειών θα το χρηματοδοτήσουν οι φορολογούμενοι, οι εργαζόμενοι κυρίω, οι οποίοι υποχρεούνται να χρηματοδοτήσουν την κερδοσκοπία των μεγάλων επενδυτών. Επιπλέον, Πολλέ φορές χάνουν και τη δουλειά τους. Και να προσθέσω και δύο ακόμα ερωτήσει. Πρώτον, και πάλι σε σχέση με την Αβέγκοα και σε ό,τι αφορά τα κριτήρια με τα οποία χορηγούνται οι πιστώσεις φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δρά σαν ένας ε, ακόμα κερδοσκοπικός ε, επενδυτής. Όμως θα μπορούσε να δράσει διαφορετικά, συνδέοντας τις πιστώσεις με τη δημιουργία ενός κοινωνικού μοντέλου επιχειρήσεων. Ε, ως ελάχιστο θα έπρεπε οι επιχειρήσεις ε, να ενισχύουν και να προωθούν την ενημέρωση και τη συμμετοχή των εργαζομένων αν είναι να λαμβάνουν χρηματοδότηση. Αυτό θα βελτίωνε πολύ την οικονομική διαχείριση και την κοινωνική συνεισφορά των επιχειρήσεων στις οποίες επενδύουμε. Το έχετε σκεφτεί αυτό. Τρίτο, τέλος, δεύτερη γενική ερώτηση. Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση που υποτίθεται το πρόγραμμα Juncker ε, θα έδινε στις κερδοσκοπικές ενεργειακές ε, ή ε, επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεταφορών. Θα ήθελα να σα ρωτήσω το εξή. Ε, έχετε αξιολογήσει τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν να έχουν τα ίδια κονδύλια αν είχε υποστηριχθεί ε, απευθείας η παραδοσιακή βιομηχανική πολιτική ή κρατικές επενδύσεις. Με αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βελτίωνε την ανταγωνιστικότητα κατευθείαν και όχι ο ιδιωτικό τομέα. Αυτό το θεωρούμε απαραίτητο για την βελτίωση της, ε, της περιφερειακής συνοχής ε, ε, και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και επίσης για την πρόθεση του κοινωνικού μοντέλου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος νομίζω είναι Το 2012 παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα εκκίνηση οικονομίας μέσω των επενδύσεων, τα ποσά. Αυτό το πρόγραμμα το είχαν ετοιμάσει οι μεγάλες δημόσιες τράπεζες και είχε παρουσιαστεί από τον κύριο Μπασανίνη το 2012 ε, με τον κύριο Μόντι Παρόν. 500 εκατομμύρια ήταν τα ποσά. Από πού θα προερχόταν? Θα ήταν πίστοση της Κεντρικής Τράπεζας ήταν ένα quantitative easing, μια δημοσιονομική χαλάρωση, μια ποσοτική χαλάρωση. Η ενέργεια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι μεταφορές λοιπά θα υποφελούνταν. η λειτουργία. Θα ήταν εντελώς διαφορετική. Είχαμε στο μυαλό μας να εξορροπήσουμε τις ε, διαρθωτικά ελληματικές χώρες. Θα δημιουργούσαμε δηλαδή μια εταιρεία επενδύσεων που θα βασιζόταν στις τράπεζες, τις δημόσιες τράπεζες, τις εθνικές δημόσιες τράπεζες για να προσανατολίσει την οικονομία σε αυτούς τους τομείς που σας ανέφερα και να δημιουργήσει νέα έργα. Οι χώρες ήταν φυσικά οι ελληματικές, διαφορετικά ελληματικές χώρες. Η λειτουργία θα ήταν αποκεντρωμένη, η οργάνωση θα ήταν κεντρική, το πώς θα διαχειριζόμασταν δηλαδή, τα έργα, πώς θα τα προετοιμάζαμε και είχαμε ζητήσει εκείνη την εποχή στο KF W να μας βοηθήσει να επιλέξουμε έργα. Αλλά δεν μας δόθηκε απάντηση. Δυστυχώς όμως αυτό το έργο δεν μακροημέρευσε. Γιατί δεν χρησιμοποίησαμε αυτά τα οικονομικά, τα νέα οικονομικά μέσα. Νομίζω ότι το πρόγραμμα Juncker έχει κάποιες δυσκολίες. Αυτές οι δυσκολίες οφείλονται στο ότι όταν μας δίνεται εγγύησεις για να κάνουμε μόχλευση, δεν δημιουργείται πραγματικά νέα έργα. Στην πραγματικότητα δημιουργείται μια ευκαιρία που υπήρχε ούτως ή άλλως, όντως, αλλά που δεν θα μπορέσει κατά ανάγκη να δράσει στου τομεί που έχουν πραγματική ανάγκη για να δώσουμε μια νέα όθηση στην οικονομία. Νομίζω επίσης ότι είναι εκ των όνου κάνευ για να υπάρξει μια ευρωπαϊκή μακροοικονομική ισορροπία να έχουμε εργαλεία τα οποία θα επιτρέψουν να εξισορροπήσουμε τον βορρά και τον νότο. Και δεν θα ρυθμίσω το πρόβλημα του ευρώ έτσι. Πώς δηλαδή τα πλεονάσματα του βορρά θα επενδυθούν στον νότο με τρόπο αποδοτικό. Χωρίς κάποια επενδυτική υπηρεσία ή φορέα δεν θα μπορέσετε να ρυθμίσετε ποτέ το πρόβλημα του ευρώ και το ευρώ είναι καταδικασμένο. Θα πρέπει να σκεφτείτε πώς θα μπορέσετε να επαναπροσανατολίσετε τελικά αυτό το πρόγραμμα Juncker, ούτω ώστε να χρησιμοποιήσετε σωστά τα νομισματικά μέσα. Ξεκινήσατε, αλλά πρέπει να πάτε στο τέλος αυτής της λογικής. Αυτά και σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σαρφάτερ. Μπλάνκο Λόπε είναι ο επόμενο ομιλητής. Ευχαριστώ. Από τις πληροφορίες που μας δώσατε. Αυτό το σχέδιο επενδύσεων ε, δημιούργησε θετικές προσδοκίες. Εγώ φοβάμαι όμως ότι από την προσδοκία πάμε στην απογοήτευση. Μας είπατε, ακόμα μια φορά, ποια είναι η κατάσταση. Μας είπατε ότι ο στόχος ήταν να διορθώσουμε την χαμηλή ανάπτυξη της οικονομίας, το πρόβλημα της απασχόλησης που είναι πολύ έντονο σε ορισμένες χώρες και να ε, αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή να ενισχύσουμε την ανάπτυξη, να δώσουμε νέα όθηση στην απασχόληση, να κερδίσουμε ανταγωνιστικότητα. Εγώ θα πρόσθετα και έναν άλλο στόχο. Το να διορθώσουμε την φοβερή ανάπτυξη ανισοτήτων που δημιουργούνται ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης. Εγώ όμως δεν είμαι σίγουρος ότι η διάρθρωση των έργων αυτών δεν είμαι σίγουρος ότι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στα έργα ε, χρησιμεύει για να δώσει νέα όθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία, για να υπάρξει ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και κυρίως για να διορθώσουμε το πρόβλημα της απασχόλησης, της ανεργίας που είναι πολύ έντονο στη χώρα μου, την Ισπανία και σε άλλες τέτοιες χώρες. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να σας, κάνω μια να σας υποβάλω μια πρόσκληση για να δείξετε μεγαλύτερη έτσι, προορατικότητα ως Επιτροπή, να δώσετε μεγαλύτερη όθηση. Γιατί αυτός ο στόχος είναι πολύ σημαντικός σε αυτή τη φάση, σε αυτή την περίοδο. Μην τον ξεχάσουμε. Επίσης, θα ήθελα να είσαστε πιο φιλόδοξοι, ούτω ώστε οι στόχοι που είχαμε θέσει, οι πολιτικοί αυτοί στόχοι, να τελεσφορήσουν. Επιπλέον, θα ήθελα, εάν δεν μπορείτε τώρα να μου απαντήσετε, να μου απαντήσετε αργότερα και να μου εξηγήσετε ποια θα είναι η συμμετοχή της ε, χώρας μου, της Ισπανίας, σε αυτά τα έργα. Γιατί η χώρα μου είναι ακριβώς μία από τις χώρες όπου η κρίση έπληξε με μεγάλη θρημίτητα και δημιούργησε ανεργία και αύξησε πολύ τις ανισότητες. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ε, αποτελούσε μεγάλη ελπίδα για την οικονομία μας. Και για εκείνους που φοβόντουσαν, δίσταζαν να επενδύσουν. Ήταν απολύτως απαραίτητο και αντιστοιχούσε σε σημαντικές προσδοκίες μας. Πρέπει να το στηρίξουμε λοιπόν, να το ενισχύσουμε, να το διατηρήσουμε. Όμως, Το εξή είναι πολύ σημαντικό και προκύπτει από τις συζητήσεις με τις επιχειρήσεις. Η πρόθεση και η προβολή αυτού του ταμείου. Οι επιχειρήσεις έχουν την εντύπωση ότι δεν καταλαβαίνουν πολύ καλά πάντα πώς λειτουργεί. Ε, δυσκολεύονται με τη γραφειοκρατική διαδικασία Αφενό έχουμε τι μεγάλες προσδοκίες από πολιτικής πλευράς, από την άλλη πλευρά όμως ε, οι διαδικασίε του Ταμείου είναι περίπλοκες, η πρόσβαση είναι δυσχερής. Δεδομένη και της κρίση, όλοι λέμε ότι είναι πήγον να χρησιμοποιηθεί, στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Πρόεδρου Γιονκέρ από την άλλη μεριά επικρατεί μια σχετική απογοήτευση. Θα πρέπει να βιαστούμε. Και τι σημαίνει αυτό, θα πρέπει να το δώσουμε περισσότερη δημοσιότητα στο Ταμείο, αλλά να ικανοποιήσουμε και τι προσδοκίε των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχουν πολλέ μικρομεσαίε επιχειρήσει που δεν έχουν τα μέσα, δεν έχουν τα μέτρα που χρειάζονται για να καταλάβουν αυτά που αναφέρονται στα αγγλικά, μάλιστα μόνο στο ίντερνετ. Γνωρίζουμε ότι τα αγγλικά είναι κοινή γλώσσα, αλλά μπείτε στη θέση των επιχειρηματιών εκείνων που βρίσκονται, δρούν στον κλάδο της καινοτομίας, δημιουργούν προϊόντα αλλά μπλέκουν σε αυτά τα γραφειοκρατικά γρανάζια και μάλιστα όλα εξηγούνται στα αγγλικά. Η Ευρώπη πρέπει να είναι η Ευρώπη της εγκύτητας των πολίτη. Και αυτό περνάει επίσης και μέσω της μετάφρασης σε διάφορες γλώσσες. Είναι απαραίτητο, πρέπει να γίνει. Για να βελτιώσουμε την κατανόηση και την αποτελεσματικότητα. Τέτοια απλά πράγματα μπορούν να βοηθήσουν. Αυτό ήθελα να σας πω. Μπέστε στη θέση αυτών των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Αγγέλικα Νίμπλερ. Τελευταία αλλά λιγότερο σημαντική. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήλθατε κύριε Μόλτερ, ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις που αναφέρθηκαν και από άλλους. Πόσα έργα διανέμονται στα κράτη-μέλη. Λέτε ότι έχετε έργα σε 24 κράτη-μέλη που έχουν χρηματοδοτηθεί μέχρι τώρα. Τι αναλογίες υπάρχουν εδώ και ποσοστά. Επίσης, ε, άκουσα ότι υπάρχουν 53 ε, έργα, αυτό το είδα από την ιστοσελίδα σας, στην Ανατολική Ευρώπη, Πολωνία, Κροατία από ένα, στη Σλοβακία ένα, είναι λίγα. Ε, ίσως θα έπρεπε να δούμε αυτή την κλίδα κατανομής. Δεύτερο, ψηφιακή, ψηφιακές υποδομές που αναφέρατε. Η ζήτηση δεν είναι μεγάλη για χρηματοδότηση. Αυτό πώς εξηγείται Κανονικά θα έπρεπε να ισχύει, ειδικά σε αυτόν τον τομέα, λόγω των εξελίξεων, μεγάλη ζήτηση. Τρίτον, με ενδιαφέρει προσωπικά, ε, εσείς ε, μετά την πρώτη, τους πρώτους μήνες λειτουργίας βλέπετε ότι οι πιθανοί επενδυτές έρχονται σε εσά ή πρέπει να κάνετε εσείς μεγάλη διαφήμιση και προωθητική ε, στρατηγική. Ευχαριστώ πολύ. Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση στο τέλος, εις ό,τι αφορά τα κεφάλαια κινδύνου που αναφέρθηκαν και στη μέση κεφαλαιοποίηση ε, εκεί. Ο συνάδελφος Τούρμες το είπε επίσης. Ε, ε έχουμε τα συστήματα εμπορίας εκπομπών επίσης και εδώ υπάρχει και ένα ταμείο καινοτομίας που εντωμεταξύ συστάθηκε. Ίσως στην αναθεώρηση θα έπρεπε τα κονδύλια που προέρχονται από εκεί να χρησιμοποιούνται 100% ενδεχομένως για έργα στον ενεργειακό τομέα που θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε τους στόχους ταχύτερα. Είναι και αυτό μία ερώτηση που ενδεχομένως θα πρέπει να συζητηθεί αλλά και να αποφασιστεί και από το Κοινοβούλιο. Ο κύριος Μόλτερερ, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις, τις εκτιμώ ιδιαίτερα γιατί μου δίνουν τη δυνατότητα να κάνω διευκρινήσεις. Ο κύριος Κάινς δεν είναι εδώ πια, αλλά αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι ότι η ανάπτυξη πάει προς μια κατεύθυνση που ευθυγραμμίζεται 100% με τον κανονισμό. Δηλαδή στο, στην ενέργεια πάει προς την κατεύθυνση ενεργειακής απόδοσης ανανεώσιμες και ανακατανομή. Στη, στο σκέλος των υποδομών δεν πιάνει μόνο την υποδομή του, του hardware αλλά μπαίνει και στην υποδομή την ψηφιακή και είναι ενδιαφέρον ότι επισέρχεται σε μεγάλο βαθμό και στην κατεύθυνση της κοινωνικής υποδομής, κοινωνική στέγη για παράδειγμα, η νοσοκομεία. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Βλέπω λοιπόν ότι έχουμε αυξανόμενη ζήτηση και στην καινοτομία, το σκέλος καινοτομίας αυτού του εγχειρήματο, αυτό σε συνδυασμό επίσης με την αυξημένη ζήτηση από την, ε, τους ιδιώτες γιατί οι ιδιωτικές εταιρείες, μέσες, μεσαίες εταιρείες κάνουν την καινοτομία. Δηλαδή η κατεύθυνση πάει καλά. Τώρα, άλλη ερώτηση. Ναι, αληθεύει ότι χρειάζεται το κομμάτι της καινοτομίας του όλου εγχειρήματο και αυτό θα πρέπει να αυξηθεί μάλιστα. Αυτό που θεωρώ σημαντικό θέμα και ίσως αυτό είναι λίγο αντιφατικό με αυτό που είπατε εσείς. Για μένα η καινοτομία δεν, είναι, δεν βασίζεται εξορισμού μόνο στην έρευνα και την ανάπτυξη. Είναι καινοτομία που προέρχεται από την παραγωγή, από την παραγωγική διαδικασία. Διότι αν κάνετε καινοτομία ε, σε στενά πλαίσια και το ορίσετε ε, στενά θα ε, βασίζεστε στη μεγάλη βιομηχανία μόνο γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι καινοτόμε, αλλά δεν μπορούν να επενδύσουν πολύ στην έρευνα οπότε πολύ εκεί. Η κατανόηση της καινοτομία λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να νοηθεί και ως συναρτωμένη με την παραγωγή. Για παράδειγμα, συνδυασμός επένδυση στην ενέργεια με την ψηφιακή ατζέντα, το ψηφιακό θεματολόγιο. Διότι αν πάτε για ενεργειακή απόδοση, αυτό συνδυάζει καλά το ενεργειακό στοιχείο, το ψηφιακό στοιχείο και τις ανάγκες έτσι της ε, πολιτικής ενέργειας. Το πίνακα ε, επιδόσεων και τα κριτήρια αυτά στα οποία στηρίζεται είναι δημόσια έχουμε εκεί μια συνολική εικόνα που βρισκόμαστε. Και ε, θα δώσω και σαφείς ενδείξεις για την έκθεση που θα ε, γίνει από την ε, Τράπεζα Επενδύσεων και με την υποστήριξή μου, χρειάζεται εδώ συμφωνία, σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συμφωνία εμπιστευτικότητας ακόμα δεν έχει γίνει. Γίνονται διαπραγματεύσει, αλλά δεν πήραμε το πράσινο φω. Και εγώ που είμαι διευθύνων σύμβουλο και δεσμεύομαι από τον κανονισμό, αυτή η ε, συμφωνία εμπιστευτικότητα είναι σημαντική για να λειτουργήσει η έκθεση. Για τι πλατφόρμε βλέπω δύο τομεί ε, ενδιαφέροντο. Το ένα είναι η ενεργειακή επάρκεια, ενεργειακή απόδοση. Διότι αν έχουμε έναν όγκο μικρότερων έργων, χρειάζεται μια δομή, ούτω ώστε αυτά να συνδέονται. Και η πλατφόρμα επενδύσεων είναι μία. Έχουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ήδη στη Γαλλία, όπου λειτουργούν καλά τα πράγματα, η εμπειρία είναι εξαιρετική και θα μπορούσε να βρει μιμητές και αλλού, ε, από άλλους ε, ομολόγους. Και η δεύτερη βασική προτεραιότητα ε, είναι η ευρεία ζώνη. Ενδεχομένως εδώ θα πρέπει να συνδυαστούν όλα τα ε, έργα σε μια μεγαλύτερη υποδομή. Πολλά μπορούν να γίνουν εδώ, πολλά βελτιωτικά. Στη χώρα που ξέρω καλύτερα όλοι συμφωνούν ότι υπάρχει ζήτηση 5-7 δις και η κυβέρνηση ακόμα έχει βάλει χρήματα για να ε, προσελκύσει επενδύσεις. Αλλά θα πρέπει όλα αυτά να συνδυαστούν. Και βεβαίως εδώ παίζει ρόλο και ίσως ε, δεν βοηθάει εδώ η ομοσπονδιακή δομή. Αυτό ισχύει και για την Αυστρία και για τη χώρα σας στη Γερμανία. Οι πλατφόρμες είναι κλειδί λοιπόν. Κύριε Τούρμες, η το εθνική υποστήριξη ναι, τα 20 συν είναι για την ε, συμβουλευτική εφαρμογή που τρέχει επιτυχώς. Πήραμε πάρα, πολλές, ε, πάρα πολλά αιτήματα, αυξήθηκαν πολύ τα αιτήματα, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι δεν είναι τόσο από το δημόσιο τομέα, γιατί αρχικά κάθε θεωρούσαμε ότι θα έρθουν από το δημόσιο τομέα. Όχι, προέρχονται τα αιτήματα από τον ιδιωτικό τομέα. Μετά, το πώς θα δομήσουμε και θα συνδέσουμε τις επενδυτικές πλατφόρμες και τρίτον είναι σημαντικό ότι πάμε προς μια κατεύθυνση του πώς θα ε, δομήσουμε τη χρηματοδότηση και τα προγράμματα ΣΔΙΤ. Αυτά είναι τα τρία. Έχουμε εμπειρία και όταν λέω εμείς ε, τυπικά δεν είναι σωστό. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει εμπειρία από την ε, χρήση συμβουλευτικών εφαρμογών. Έχει μια συμφωνία με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία η Τράπεζα Επενδύσεων όπου ε, το συμβουλευτικό κομμάτι και το κόστος του καλύπτεται από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Οπότε υπάρχει θετικό παράδειγμα που έχει εφαρμοστεί, αλλά περιορίζεται αυτή τη στιγμή μόνο σε αυτά που σας είπα. Τώρα, οι ανατολικές χώρες, γιατί δεν ε, έχουν πολλά έργα ακόμα. Δύο εξηγήσεις εδώ. Καταρχήν, ναι, είναι σωστό ότι θέλουμε τις τεχνικές συμβουλές του ώστε να φτιαχτούν τα έργα και να σχεδιαστούν, αλλά θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχει κι άλλος ένας λόγος. Δηλαδή ε, αναφέρουμε στην οικονομική δομή, στη δομή της οικονομίας των χωρών. Αν δούμε ας πούμε τη Δυτική Ευρώπη όπου έχουμε πολλές ε, και συγκρίνεται με τις χώρες όπου η, οικονομική, δομή της οικονομίας δεν είναι τόσο προχωρημένη, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα, ε, μια εξήγηση και το, η τρίτη εξήγηση που έχει να κάνει με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι η ικανότητα της διακυβέρνησης στον τομέα της διαχείρισης. Τώρα για τον πολλαπλασιαστή, μια διευκρίνηση. Αυτό που βλέπετε είναι ο εξωτερικός πολλαπλασιαστής μόνο το 1 προς 15 έχει να κάνει και με τον εσωτερικό και τον εξωτερικό πολλαπλασιαστή. Αυτό που πρέπει να προσθέσουμε είναι λοιπόν τον εσωτερικό πολλαπλασιαστή που πάει από τις εγγύσεις στα 10,5 δις ε, χρηματοοικονομικά μέσα. Αν τα συνδυάσετε αυτά, τα προσθέσετε, μπορείτε να πείτε ότι είμαστε εντάξει με τον ε, ε, πολλαπλασιαστή που είχαμε προβλέψει. Ο πολλαπλασιαστή δεν ισχύει μόνο για ένα έργο όμως, αλλά για το ε, χαρτοφυλάκιο του όλου εγχειρήματο του Ταμείου. Κύριε Μπέκαρ, να σας δώσω μια ένδειξη για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και αυτό είναι καινούριο για την τράπεζα αυτή. Ε, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της ε, τράπεζας έχει κάποιες ενδείξεις για τις λεγόμενες ειδικέ δραστηριότητες. Δηλαδή 2 με 4 δις από τα 72 συνολικού ε, τώρα, το ποσό για φέτος έχει αυξηθεί στα 20 με 25 Δηλαδή εδώ αλλάζουν σημαντικά οι όροι του παιχνιδιού, έχουμε λιγότερο από 10% και πάει προς την κατεύθυνση του ενός τρίτου. Και αυτό είναι σημαντικό. Και αναφέρεται στις ερωτήσεις σας. Τώρα, οι ε, ε, επιλογές για προσέλκυση ενδιαφερομένων, ε, δύο βασικές, ό,τι είναι δυνατόν να γίνει γύρω από τις επενδυτικές πλατφόρμες οι οποίες εξορισμού προσελκύουν ιδιωτικό κεφάλαιο και δεύτερον θα πρέπει να έχουμε δομημένη χρηματοδότηση στις υποδομές. Αν έχουμε ένα πρόγραμμα ΣΔΙΤ εξορισμού, αυτό προσελκύει ιδιωτικό κεφάλαιο. Και το τρίτο στοιχείο βέβαια είναι να έχουμε το Ταμείο των Ταμείων Fund of Fund ιδιαίτερα στη, στα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου ε, και να δίνονται κίνητρα από την τράπεζα και το Ταμείο αφού τα περισσότερα χρήματα προέρχονται από τους ιδιώτες. Ε, τα ίδια κεφάλαια θα πρέπει να προσεχθούν, να αναπτυχθούν η έμεση, ε, τα έμεσα ε, ναι, ε, ίδια κεφάλαια συζητούνται, γίνεται μια συζήτηση και για άμεσα ίδια κεφάλαια. Αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί γιατί τα άμεσα ίδια κεφάλαια είναι καινούργια και για την Τράπεζα Επενδύσεων και δεν είναι εύκολο να τα προχωρήσουμε γιατί χρειάζονται προετοιμασίες και ιδιαίτερες ικανότητες. Εκεί που θα διαφωνήσω μαζί σας είναι όταν λέτε ότι μία εγγύηση στις τράπεζε από την Τράπεζα και το Ταμείο Επενδύσεων ε, είναι ε, ε, χρηματοδότηση εμέσως. Η ε, ε, ελάφρυνση είναι ένας τρόπος για να αυξήσουμε τη δανειοδοτική δυνατότητα των τραπεζών, γιατί η προϋπόθεση για την ε, ελάφρυνση ε, κεφαλαιακή είναι η πρόσθετη χρηματοδότηση. Αλλιώς δεν θα μπορούσαν να έχουν ε, κεφαλαιακή ελάφρυνση οι τράπεζες. Άρα λοιπόν δεν είναι χρηματοδότηση των τραπεζών. Τι κάνει η, τράπε... η, η ΕΚΤ, η Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δίνει ρευστότητα ε, πιέζει τις εμπορικές τράπεζες ε, για, ε, προς την κατεύθυνση του δανεισμού. Εδώ μεταξύ οι τράπεζες έχουν και, και περιορισμούς και αυτό δεν τις διευκολύνει. τα μέσα λοιπόν κεφαλαϊκής ελάφρυνσης είναι μία δυνατότητα αύξησης της δανειοδοτικής ικανότητας, ιδιαίτερα προς τις ΜΜΕ από τις εμπορικές τράπεζες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Για την Ισπανία έχουμε πολλά έργα εκεί, αυτό είναι βέβαιο. Η Σναμπεγκόα, την ξέρουμε, είναι μια εταιρεία υπό ανά ε, ε, η τράπεζα περιμένει την ανασυγκρότηση της εταιρεία για να προχωρήσει στην εκταμίευση. Ακόμα δεν έχει γίνει εκταμίευση. Έτσι έχει το θέμα. Τώρα, για να γίνει μια σύγκριση μεταξύ ε, παραδοσιακής ε, χρηματοδότησης υποδομών και χρηματοδότησης με βάση ε, μια σύμπραξη ΣΔΙΤ, αυτό είναι διαφορετικό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το θέμα δεν είναι να συγκρίνουμε την δομημένη χρηματοδότηση με την παραδοσιακή. Το θέμα είναι διαφορετικό τώρα. Δηλαδή, επενδύσεις γίνονται χωρίς δομημένη χρηματοδότηση, γιατί έχουμε περιορισμένες δυνατότητες ε, του δημοσίου τομέα. Βλέπουμε ότι οι εταιρείες κάνουν ακριβώς τη σύγκριση αυτή, αλλά και με άλλες πηγές χρηματοδότηση. Και το «Ιρισδίτε» δεν είναι θέμα ιδεολογικό, είναι μια ρεαλιστικότατη προσέγγιση. Αν αυτό είναι το μέσον για να γίνουν επενδύσεις, ας το χρησιμοποιήσουμε. Αν θέλουμε να κάνουμε ιδεολογική συζήτηση για τις επενδύσεις, ε, τότε ε, απλά επενδύσεις δεν θα γίνουν άμα θεωρητικολογούμε. Εγώ αυτό ξέρω να πω. Κύριε Σαρφχάουζεν, ε, για την επενδυτική πλατφόρμα και τα NPPs. Εδώ και μερικές εβδομάδες υπάρχει ένα έγγραφο στρατηγικής NPPs ε, και προσέγγιση έτσι. Μπορούμε να, μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα. Ε, η τράπεζα ετοιμάζει τώρα και χρησιμοποιεί έργα για τη συνεργασία με την NPP. Η συνεργασία και το εύρος με την NPP είναι μεγάλη. Υπάρχει μια εκδήλωση ε, που προγραμματίζεται για την επόμενη, τις επόμενες 6-8 εβδομάδες. NPP συζήτηση θα γίνει και εδώ στην Επιτροπή Προϋπολογισμών όπου είναι αυτό ένα θέμα και είμαστε βέβαιοι ότι το προϊόν, ε, το, η εργαλειοθήκη στις NPP θα αυξήσει τις δυνατότητές τους. Τώρα, νομίζω ότι καλύπτουν, καλύπτει ο κανονισμός τις ανάγκες των τομέων. Ε, είναι αρκετά ευρέως διατυπωμένος ο κανονισμός. Κατανοητό. Από την άλλη έχουμε σαφή ένδειξη ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε παράλληλα με τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ενέργεια, ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση κλπ. Και το εύση δεν είναι πανάκια. για να λύσει όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Και αν είναι υπερβολικές οι προσδοκίες από το έτσε, δηλαδή να πιάσει όλο το θέμα της συνοχής και να το λύσει, να <clears throat> ξεκαθαρίσει όλα τα, όλες τις άλλες ανάγκες για τις διαφορετικές ε, μετακμίσεις, ε, τότε θα μας παραφορτώσετε. Το έτσε δεν είναι πανάκια είναι ένα μέσον και γι' αυτό είπα στην εισαγωγή μου ότι το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη συνίσταται σε τρεις πυλώνες και όχι σε μία. Σένια Λόπες, ε, Ελπίδα και Ματέωση. Χθε είχαμε μια μεγάλη εκδήλωση, για παράδειγμα, εδώ στις Βρυξέλλες. Μου φαίνεται 600 επιχειρηματίες ήρθαν. Και πρέπει να σας πω ότι το κλίμα στη χθεσινή συνεδρίαση ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και τι είπαν οι επιχειρηματίες, ιδιαίτερα οι μικρότεροι. Είπαν ότι αυτό είναι ένα μέσο που μας δίνει προοπτική. Και περί αυτού πρόκειται. Είναι ένα μέσο που δίνει προοπτική επενδύσεων και αυξάνει την ανταγωνιστικότητα, συμβάλλει δε επίσης και στην άμβληση των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας και την πολύ επικίνδυνη κατάσταση στην αγορά εργασίας. Ε, Επιβεβαιώνω λοιπόν και νομίζω όλοι μπορούμε ε, να επιβεβαιώσουμε ότι αυτό, και αυτή είναι και η κοινή γνώμη, ότι αυτό είναι ένα μέσο που δίνει ελπίδα. Κυρία Γκροστέτ, μάλιστα, πρέπει να γίνει πρόθεση, πρέπει να το, το διαφημίσουμε αυτό το μέσο. Και τώρα κάνουμε πολλά ταξίδια, πολλά, πάμπολα, από πρωτεύουσα σε πρωτεύουσα. Και πάμε και σε περιφέρειες γιατί πολλά από αυτά τα έργα είναι περιφερειακά. Χθε, για παράδειγμα, ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που έγινε και ίσως μπορεί να το εξετάσουν και άλλες χώρες. Η χώρα, η δικιά σας, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Έχουν ορίσει έναν λεγόμενο επίτροπο για επενδύσεις. Είναι δηλαδή κάποιος που ασχολείται ειδικά με αυτό το θέμα. Το έργο του είναι να προσελκύσει και να προσεγγίσει εταιρείες δημόσιες και ιδιωτικές και να είναι ένας σύνδεσμος μεταξύ αυτών και των αναγκών τους. Και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Άριστο παράδειγμα και βέβαια και αυτό το Ταμείο για την Κοινωνική Στέγαση και αυτό το έργο στην Γαλλία ήρθε σε επαφή με το ΕΤΣΕ, με το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, με αυτόν τον διευκολυντή αν θέλετε, με αυτόν τον ενδιάμεσο που έχει οριστεί. Ε, για την διοίκηση. Έχετε δίκιο από τη μια, αλλά από την άλλη πρέπει να ξεκαθαρίσω και κάτι ακόμα. Ο κανονισμός που εγκρίνατε δεν ε, μειώνει το βάρος διότι όταν πρόκειται για τις ανάγκες υποβολής εκθέσεων που σας ενδιαφέρει πολύ, ε, αυτές οι ανάγκες είναι κομμάτι της σύμβασης με τον συμβαλόμενο. Γιατί αλλιώ πώ θα γίνει σωστή έκθεση. Πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία λοιπόν μεταξύ όλων των ε, αναγκών, ε, συμμόρφωση, ε, δημοσίων συμβάσεων κλπ. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προσπαθεί να το κάνει αυτό. Αλλά έχετε δίκιο. Αυτό είναι ένα θέμα που πάντα ασκεί πιέσει στην τράπεζά μας. Τώρα, τα περιφερειακά γραφεία ανοίγουν σιγά-σιγά στις παλιές ε, πρωτεύουσες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βοηθούν πολύ. Κυρία Νίμπλερ, έχουμε 54 έργα, αλλά όχι και στα 28 κράτη-μέλη. Είναι 14 από τα, σε 13-14 από τα 28. Και αυτό είναι και αυτό που είπε ο κύριος Τούρμες, ότι πρέπει να αυξήσουμε την ικανότητα παρα... ανταπόκρισης σε ό,τι αφορά τα έργα υποδομής και τα ιδιωτικά έργα σε αυτές τις χώρες. Τα άλλα καλύπτονται από το, ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Επενδύσεων και εδώ ε, για να πω και κάτι θετικό, την επόμενη εβδομάδα θα καλύπτουμε 25 κράτη-μέλη. Το, η δραστηριότητα του Ταμείου Επενδύσεων ε, σε αυτές τις χώρες είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντική, γιατί απευθύνονται στις ΜΜΕ που είναι η ραχοκοκαλιά εδώ. Πρέπει λοιπόν να λαμβάνονται οι αποφάσεις ε, με βάση τη σημασία του έργου. Εμείς δρούμε ως όμιλος, δηλαδή και τράπεζα και ε, το κομμάτι της ε, έρευνας και καινοτομίας. Ε, σίγουρα είναι μόνιμη πρόκληση το πρόγραμμα για τους πρεσβευτές του ΕΤΣΕ, γιατί και καλό είναι να συμμετέχετε γιατί ξέρετε επιτοπίως την κατάσταση και αν ε, τύχουμε κάποιας υποστήριξης θα ήταν προς το συμφέρον όλων. Πάουλ Ρούμπικ για τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου. Ναι, υπάρχει αυξημένη ζήτηση ε, και τέτοιων κεφαλαίων, το βλέπουμε στην αγορά. Ε, επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητεί εντατικά τώρα για να δημιουργήσει ένα fund of fund για κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να προσελκύσει και ε, επενδυτές από το εξωτερικό που καμιά φορά έχουν πρόβλημα με τα μικρά ταμεία περιφερειακής βάσης. Γι' αυτό θέλουμε να έχουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Fund of Funds και ε, εδώ θα αξιοποιηθεί και η εμπειρία του Ταμείου Επενδύσεων. Ε, τέτοιο, αν υπάρχουν ιδέες για την αξιοποίηση ενός τέτοιου Ταμείου Επενδυτικών Κεφαλαίων, ε, κεφαλαίων υπαχειρηματικού κινδύνου, είναι ευπρόσδεκτες. Επίσης, το ε, περιβάλλον, το περιβάλλον των νεοφιών επιχειρήσεων στην Ευρώπη δεν είναι τόσο δυσμενές πλέον. Εμείς ε, θέλουμε να αναβαθμίσουμε τις ε, νεοφυείς, αν έχουν επιτυχία, κλείνοντας το δημοσιονομικό κενό που υπάρχει στη δεύτερη φάση ανάπτυξης αυτών των νεοφυών. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και είμαι έτοιμος να ξαναέρθω στην Επιτροπή σας αν με προσκαλέσετε. Äh, Ο Κλοντ, δύο, λεπτάκια, μια παρατήρηση ακόμη. Είχα μια ερώτηση ε, από την ε, για την Κομισιόν, οπότε πώς θα μπορούσαμε να, να πάρουμε μια πόνση την απαντήσεις τη πήραμε, η Κομισιόν θα επανέλθει προσωπικά σε σένα και θα σου δώσει λεπτομερείς εξηγήσεις. Έχει καλώς. Και έτσι... Α, κάποιος ακόμα ζητεί το λόγο. Ορίστε. Για το σχόλιο που έκανε ο Γενικό κύριος Διευθυντής. Ε, δύο λογάκια μόνο. Ε, ότι πρέπει να είμαστε πρέσβης. Δεν το έχουμε κάνει ως τώρα. Πρέσβης ε, προκειμένου να προωθήσουμε ε, ε, κάποιο project. Το έχουμε κάνει μία φορά, αλλά περιμένουμε τρεις μήνες απάντηση αυτή τη στιγμή. Οπότε πραγματικά είναι πολύ περίπλοκη η διαδικασία. Okay. Πέστε μου για ποιο project μιλάτε. Πολύ ευχαριστώ. Να, το, να προωθήσω το σχόλιο σας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Äh, Ευχαριστώ πολύ. Είναι σε καλά χέρια το έτσι. Βέβαια είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τακτικές επαφές, γιατί ε, εμείς ως Επιτροπή Βιομηχανίας θέλουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση, να στηρίξουμε και τα έργα, ε, να γίνουμε ευχαρίστως πρεσβευτές του έτσι στις χώρες, mail, στις χώρες καταγωγής μας. Ευχαριστώ πολύ και ή από τώρα αναγγέλλω ότι θα έρθει και επόμενη πρόσκληση ε, για να παρευρεθείτε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Äh, Καλώς. Πάμε στο επόμενο. Μετεκλογική αναθεώρηση 2014-2020 το Κοινοβούλιο ήδη από τώρα προσπαθεί να παρουσιάσει τις δομές σε μια πρωτοβουλία. Ο συντάκτης μας είναι ο Γιάννος Λεβαντόφσκι, πρώην Επίτροπος. Είναι πολύ σημαντικό, ε, πιστεύω, μέχρι το 2030 να έχουμε ε, επιτύχει το 20% αύξηση της παραγωγής στην Ευρώπη και βεβαίως πολλές καινοτομίες. Θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Λεβαντόφσκι για να μας παρουσιάσει τις απόψεις τους. Ο κανόνας, το άρθρο 53 ε, προβλέπει ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών είναι επί της ουσίας. Μέχρι το τέλος του 2016 θα πρέπει να υποβληθούν οι προτάσεις για την αναθεώρηση. Εμείς ε, έχουμε τα προγράμματα Γαλιλαίο, Πέρνικου στο ΣΕΦ, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ίσως το Εράσμους για νέους ε, επιχειρηματίες, επιχειρηματίες μεταναστών. Είναι πολλά τα έργα και πολλή δουλειά. Γιάννους, το πιο σωστό είναι να παρουσιάσουμε έγκαιρα τις απόψεις μας. Ε, παρακαλώ, έχεις το λόγο για να μας παρουσιάσει το θέμα. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Ιτερε θα πρέπει να απεικονίζει την ευαισθησία που δείχνει η Επιτροπή μας στο θέμα αυτό. Πρέπει να μην ξεχνάμε τι πρέπει να αναθεωρηθεί, που είναι το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι δημοσιονομικές προοπτικές που είναι χαμηλότερες από τις προηγούμενες. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Συνήθως ε, αυξάνουν οι ευρωπαϊκοί προπολογισμοί. Λόγω όμως των ισχυρών πιέσεων και από τον κύριο Κάμερον και λόγω της δημοσιονομικής εξυγίανσης στα κράτη-μέλη, οι δημοσιονομικές προοπτικές 2014-2020 συρρυκνώθηκαν σε σχέση με τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές του 2007-2014 κατά 30 δις. Υπάρχει λοιπόν ε, ένα χάσμα ανάμεσα στους πόρους που διαθέτουμε και στις ε, πολύ περισσότερες ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε μια πραγματική εκβάθρο αναθεώρηση, όχι μια επιφανειακή επανεξέταση. Και συνεχεία μια νομοθετική αναθεώρηση των συνεχόμενων δημοσιονομικών προοπτικών που τρέχουμε μέχρι το 20. Μην ξεχνάτε ότι και το εξωτερικό περιβάλλον άλλαξε άρδιν. Έχουμε νέα έργα όπως το ΕΦΣΙ που συζητήσαμε τον κύριο Μόρτερεν, καθώς και νέες απαιτήσεις, νέες προκλήσεις, κυρίως διαχείριση της μετανάστευσης και της α, πολιτικής των προσφύγων. Όλοι αυτοί οι λόγοι απαιτούν μία εκβάθρον αναθεώρηση και όχι μία επανεξέταση. Και η δική μας Επιτροπή ξέρει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει εις των δικών μας προγραμμάτων, του Ορίζοντα 2020, του Κόσμε, της έρευνας εν γέννη. Και αυτό ακριβώς αναφέρει και το σχέδιο γνωμοδότησής μου. Αυτά που πήρανε από το ΕΦΣΥ θα πρέπει να ανακτηθούν στο, στην τρέχουσα περίοδο μέχρι το 2020. Αυτή την ευαισθησία δείχνει η Επιτροπή Ήτρε οι προτεραιότητές μας που έχουν εκφραστεί και έχουν συμφωνηθεί στα πλαίσια του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου και που ισχύουν όπως ισχύουν και οι προτεραιότητε του ΕΦΣΥ. Αν έχουμε λιγότερα λεφτά, λόγω ε, αυτού του Ταμείου Εγγυήσεων και τη εκταμείευση που γίνεται από αυτό, θα πρέπει να ανακτηθεί αργότερα. Φυσικά, αυτό που συζητήσαμε με τον κύριο Μόντερεν είναι η ανάγκη για μεγαλύτερη συνέχεια μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων του ΕΦΣΙ, των διαρθωτικών ταμείων, του Horizon, του COSME και όλων των προγραμμάτων της ΉΤΡΕ. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επίσης. Χρειάζονται καλύτερη χρηματοδότηση και αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό και η Κομισιόν θα πρέπει να το κάνει είναι μέχρι το τέλος του 2016 να κάνει μια πρόταση αναθεώρησης. Επίσης θα πρέπει να δούμε και σε τι φάση εφαρμογής είμαστε. Έχουμε καθυστερήσει. Θα πρέπει να κρίνουμε τις επιδόσεις, θα πρέπει να δούμε τις ε, μελλοντικές προοπτικές με βάση τις σημερινές επιδόσεις. Άλλοι ξέρουν ότι έχουμε ήδη καθυστερήσει. Η συμφωνία έγινε καθυστερημένα, ε, οι διαπραγματεύσεις καθυστέρησαν ε, και ήδη ε, έχουν πληρωθεί ένα δισεκατομμύριο λιγότερο ε, σε πληρωμές πέρυσι. για τα πολιετή ε, προγράμματα. Όταν βλέπουμε τη φάση εφαρμογής, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα είναι καθυστερημένα. Καθυστερεί η συμφωνία, καθυστέρησε η εφαρμογή και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αυτό είναι το περιεχόμενο ουσιαστικά της ε, γνωμοδότησής μου. Ευχαριστώ. Οι δομές έχουν αλλάξει πολύ, οπότε το Κοινοβούλιο θα πρέπει έγκαιρα να γνωρίζει τι συμβαίνει, πώς θα εφαρμοστούν τα προγράμματα Κυρία Μούρη. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Λεβαντόφσκι. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τα όσα ανέφερε. Είναι κοινός πάνω για όλη μας την Επιτροπή. Λαμβάνοντας δε υπόψη και την συζήτηση που είχαμε ε, πριν από λίγο για, τον έτσι, για το έτσε. Ε, επηρεάζει και το τμήμα αυτό του προπολογισμού. Υπάρχουν και κοινέ ε, προτεραιότητες με το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, αλλά τα πράγματα γίνονται με πολύ διαφορετικό τρόπο, διαφορετικό τύπο χρηματοδότηση, δηλαδή και θα πρέπει να τις υπογραμμίσουμε αυτές τις διαφορές, να τις αναγνωρίσουμε. Οι μειώσεις που έγιναν εξαιτία του ΕΤΣΕ θα πρέπει να ανακτηθούν, είναι προτεραιότητα. Επίσης, συμφωνώ με την, το θέμα για την καλή διαχείριση του ε, ορίζοντα, ορίζοντα 2020 και να αποφύγουμε την υστέρηση των πληρωμών που μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο. Μετά, ε, η κυκλική οικονομία, βιομηχανική πολιτική και η ε, ενεργειακή ένωση πρέπει να είναι προτεραιότητές μας και τέλος ο προπολογισμό με βάση τα αποτελέσματα ε, και ο ορισμός αυτής της έννοιας ε, θα πρέπει να δώσουμε και εμείς την ερμηνεία μας για το τι πρέπει να σημαίνει ένας τέτοιος προπολογισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Νουνχάουζεν από του Φιλελευθέρου εξ του κυρίου Φιλίπ Τεμπάκερ, ο οποίος είναι εισηγητής ε, για τα εγχειρίδια, ε, οπότε είναι στην Επιτροπή Έκων αυτή τη στιγμή. Αναφέρει τα εξή, συνάδελφοι. Όπως και οι προηγούμενοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λεβαντόφσκι για αυτή την ε, έκθεση. Λαμβάνει σίγουρα υπόψη τα περισσότερα από τα πράγματα που είναι σημαντικά για μένα και την ομάδα μου ε, με ικανοποιεί το κείμενο γιατί αναφέρει σαφώς ότι πρέπει και θα αποδώσουμε την απαραίτητη σημασία στην αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Οι συζητήσεις, δημοσιονομικές συζητήσεις για το επταετές ε, είναι μακρές και δύσκολες, οπότε όταν γίνονται μακρο, μακρόπνοες αλλαγές θα πρέπει να προσπαθούμε να προσπίσουμε τα συμφέροντά μας και να διασφαλίσουμε ότι θα εξασφαλίζεται πολιτική ισορροπία. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της έκθεσης, της γνωμοδότησης, με ικανοποιεί πολύ. Αναφέρεται σαφώς την ε, διαφορά ανάμεσα στους, ε, στο στόχο του ορίζοντα 2020 και το έτσε. Ο Επίτροπος κ. Κατάινεν τον περασμένο μήνα σε αυτή την Επιτροπή ήταν πολύ σαφή. Τα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΤΣΕ είναι τελείω διαφορετικά, πολύ διαφορετικά από αυτά τα οποία θα χρηματοδοτούσε ο Οριζόντα 2020. Αυτό καθιστά ακόμα πιο σαφή τη στάση μας. Ε, είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για την βασική έρευνα, τα κονδύλια του ορίζοντα 2020 να ανακτηθούν. Το ίδιο ε, ε, προφανώς αφορά και τα, τα κονδύλια του έτσε. Ε, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στι μικρομεσαίε επιχειρήσει ε, και κυρίω ε, στο τι χρηματοδότηση χρειάζονται περισσότερο σήμερα, αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, χρηματοδότηση κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι επενδύσεις με ψηλότερο κίνδυνο αλλά και υψηλότερη απόδοση θα λάβουν την απαραίτητη χρηματοδότηση προκειμένου να αναπτυχθούν θα υποβάλω και κάποιες τροπολογίες για αυτό το θέμα. Τελειώνω λέγοντας μία ακόμα φορά ότι η νομοδότησία είναι πολύ καλή βάση συζήτηση και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος της διαδικασίας θα υποβάλουμε μία φιλόδοξη και ισορροπημένη ε, γνωμοδότηση στους ε, συναδέλφους της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Ο κ. Μαραγκάλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συνεργαστούμε πολύ καλά με τον κύριο Λεβαντόφσκι για να προσπίσουμε τα συμφέροντα της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Συμφωνώ με τον πρώτο στόχο. Νομίζω ότι συμφωνούν όλοι με αυτό το στόχο και με όλες οι επιτροπές. Μιλάμε για μια αναθεώρηση, κάτι το οποίο σημαίνει αλλαγή, προσαρμογή, νέες προτεραιότητες, καινούριου στόχου κλπ. Η υπόσχεση για την προστασία του ορίζοντα 2020, η δέσμευση για την προστασία, θα πρέπει να είναι το ελάχιστο σημείο αφετηρίας. Δεν μπορούμε όμως να θεωρήσουμε ότι είναι κερδισμένη μάχη. Ε, θα έπρεπε ε, δυστυχώς να είναι το σημείο αφετηρίας, αλλά δεν είναι. Ε, δεν θα έπρεπε να είναι η μεγάλη μα μάχη, αλλά δυστυχώ είναι Το ελεγκτικό συμβούλιο βέβαια, συνέδριο, είπε ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν επαρκεί ενδεχομένω για να καλύψει την στρατηγική 2020. Ε, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα αυτά δύο, ένα χάσμα και θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να το καλύψουμε, να ορίσουμε ε, κριτήρια για περικοπές προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι. Ο γενικός στόχος θα έπρεπε να είναι η αύξηση των οροφών για τις, ε, ε για τις πιστώσεις αλλά και για τις πληρωμές. Θα πρέπει να το κάνουμε αυτό για να, έχουμε, για να αυξήσουμε την ευελιξία την οποία έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια. Και θα πρέπει να έχουμε ευελιξία γιατί η κατάσταση είναι ρευστή. Τρίτον, υφίσταται ο κίνδυνος σε αυτή την αναθεώρηση ε, με τους καινούριους στόχους, με τις καινούριες προτεραιότητες να προκύψουν καινούριες ε, ε, ανισορροπίες ε, μεταξύ των κεφαλαίων. Εμείς θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτά τα κεφάλαια, σε αυτούς τους τομείς που εμείς έχουμε περισσότερη ανάγκη. Άμι, βρισκόμαστε σε άμυλα με 12 επιτροπές αυτού του Κοινοβουλίου. Να σας πω δύο λόγια μόνο ακόμα, Πρόεδρε. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στην αναθεώρηση την ε, την, τους, την πλήρη εφαρμογή των, ε, των υποσχέσεων των δεσμεύσεων που λάβαμε στην COP21 χωρίς ε, ε, η, χωρίς ιδεολογικές μανίες και τρίτον θα πρέπει να περάσουμε πιο πολύ στα δάνεια και λιγότερο σε δωρεάν βοήθεια. Ε, όμως ε, προσοχή, μην πάρουμε από τον προπολισμό κεφάλαια και τα περάσουμε σε άλλα μέσα ε, τα οποία δεν θα μας χρησιμεύσουν. Äh, äh, Κυρία Σακοράφα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λεβαντόφσκι για την αρχική προσεκτική και περιεκτική προσέγγιση του κρίσιμου ζητήματος της ενδιάμεσης επανεξέτασης λειτουργίας και εφαρμογής καθώς και της μετακλογική αναθεώρησης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Δύο είναι οι δέσμες θεμάτων, κατά την άποψή μου, πάνω στις οποίες καλούμαστε να πάρουμε άμεσα θέση. Η πρώτη, στην οποία και θα αναφερθώ εκτενώς, σχετίζεται με τη βελτίωση της ευελιξίας του τρέχοντος πλαισίου και την αναθεώρηση των ανώτατων ορίων του. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, το νέο πλαίσιο ήταν προϊόν μιας ταραχώδους διαπραγμάτευσης που κατέληξε σε χαμηλότερο όριο συνολικών δαπανών σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο, όπως παραδέχτηκε και ο κύριος Λεβαντόφσκι προηγουμένως στην εισήγησή του. Και αυτό έγινε παρά τις αυξημένε αρμοδιότητες που απέκτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και παρά την ε, ε, πρόσφατη διεύρυνσή τη. Η μονόπλευρη λογιστική προσέγγιση από ορισμένα κράτη-μέλη που θεωρούν τι εθνικέ συνεισφορέ έξοδο που πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο. Η σχεδόν πραξικοπηματική εισαγωγή τη αντιαναπτυξιακή και ακρεπτών νεοφιλελεύθερη έννοια τη μακροοικονομική αρεσιμότητα στην πολιτική συνοχή. Η έλλειψη γνήσιου διαλόγου για τι προτεραιότητε και η απροκάλυπτη προσπάθεια παραγωνισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την διαπραγμάτευση οδήγησαν σε μεγάλε καθυστερήσει για την επίτευξη τη συμφωνία και στην εκκίνηση τη εφαρμογή. Οι δραματικέ εξελίξει σε διεθνέ ε, κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, όπω επίση επισήμανε ο κύριο Λεβαντόφσκι και αναφέρομαι στην προσφυγική κρίση, την οξία και παρατηταμένη κρίση στην Ελλάδα και όχι μόνο, και τα τρομοκρατικά χτυπήματα, δημιουργούν από μόνε του συνθήκε για επίγουσα ανακατανομή των ήδη περιορισμένων διαρθρωτικών πόρων. Επιπλέον, η δημιουργία του εξαιρετικά αμφίβολου Ταμείου για τι Στρατηγικέ Επενδύσει έρχεται με τη σειρά τη να περικόψει παραπέρα τον αναπτυξιακό κουμπαρά και μάλιστα σε βάρος προγραμμάτων με αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία όπως είναι ο ορίζοντας και το κόσμο, ενώ δεν θα πρέπει στιγμή να λησμονούμε την βραδιφλεχή φόβα των ανεξόφλητων λογαριασμών στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Όλα τα παραπάνω οδήγησαν στην πρόορη και μαζική ενεργοποίηση του συνόλου των ειδικών μηχανισμών, εργαλείων ευελιξίας και διαδικασιών έσχατης λύσης που προβλέπονται από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, εγείροντας πλήθος ερωτημάτων για την επάρκεια των πόρων και την αποτελεσματικότητα των δράσεων σε σχέση με τις εκρηκτικές τέρακουσε ανάγκες. Είναι λοιπόν μονόδρομος η σαρωτική αναθεώρηση με γενναία αύξηση των ορίων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, χωρίς να γίνεται κάμια έκπτωση στην δημοκρατική νομιμότητα. Η δεύτερη δέσμη θεμάτων, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, έχει προδραστικό χαρακτήρα στην κατεύθυνση τη παραπέρα βελτίωση τη χρήση των διαρθρωτικών πόρων μετά το 2020. Επιγραμματικά θα αναφέρω την ανάγκη για ένα γνήσιο σύστημα ίδιων πόρων, την αντιστοίχηση τη περίοδου εφαρμογή των μελλοντικών πλαισίων με τι θητείε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή, την επικέντρωση στα αποτελέσματα, την απλούστευση των διαδικασιών, καθώς και τη συμπερίληψη κάθε δαπάνη στον ενιαίο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ολοκληρώνοντας λοιπόν την αρχική μου παρέμβαση, θα δηλώνω πρόθυμη, αλλά και για επικοδομητική συνεργασία και κάθε πρόταση που θα ενδυναμώσει τις απόψεις του τρέχοντος σχεδίου που κινούνται πάντα σε θετική κατεύθυνση, κύριε Λεβαντόφσκη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Äh, Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή μας να έχει ενίο μέτωπο και ισχυρή φωνή σχετικά με την έκθεση πρωτοβουλίας. Πρέπει λοιπόν οι προτάσεις να είναι εστιασμένες, άρα και εφαρμοστέ, ε, εφαρμόσιμες. Έχουμε και την Κομισιόν εδώ ο κύριος Νόνενμαν θα κάνει κάποιο σχόλιο μετά από τις ερωτήσεις, παρεμβάσεις. Εδώ ε, έχουμε βέβαια το Γαλιλαίο, το Κοπέρνικους, ε, θέματα απασχόλησης κυρίως. Ε, μπορείτε να μας κάνετε μια παρουσίαση, ε, παρέμβαση 3-4 λεπτά. Ευχαριστώ από την DG Grow. Επιβεβαιώνουμε ότι εργαζόμαστε επί αυτής της αναθεώρησης. Είμαστε σε αρχική φάση. Δεν έχουμε συμφωνήσει τη μερίσια διάταξη για την επαφή μας με το Κοινοβούλιο. Το μόνο που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι προσπαθούμε να σεβαστούμε αυτά που συμφωνήθηκαν στα προηγούμενα πολιετή δημοσιονομικά πλαίσια και να εκτελέσουμε με κάθε προτεραιότητα αυτά που συμφωνήσαμε και να κρατήσουμε αυτά τα project όπως το κόσμο, Κοπέρνικους και Γαλιλαίο. Να τα κρατήσουμε υγιή, ακέραια ε, και μακριά από αλλαγές και αστάθεια. Αλλά και η πραγματικότητα είναι αυτό που είναι, έτσι. Γίνονται πολλές συζητήσεις επίσης στο πώς θα επικοινωνήσουμε ούτως ώστε ο προϋπολογισμός να δώσει αποτελέσματα. Εργαζόμαστε εργοδός. Δεν μπορούμε να σας δώσουμε συγκεκριμένες ημερομηνίε ακόμα όμως, αλλά σίγουρα θα έρθουμε προσεχώς σε επαφή μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για το χρονοδιάγραμμα. Αυτά από πλευράς μου. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε από την αρχή έγκαιρα. Η DG Gross είναι ένας καλός εταίρος και θέλω να ευχαριστήσω κύριε Νόενμαν για την προσφορά συνεργασίας και συντονισμού. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Έχουμε εισηγητή και τον παρακαλούμε να μας πει τη γνώμη του για το... Α, να μας πει ο εισηγητής τι σκέφτεται να κάνει από εδώ και πέρα στα πλαίσια των προθεσμιών που υπάρχουν γιατί μέχρι 21 Απριλίου πρέπει να κατατεθούν οι τροπολογίες, μάλλον στις 24 Μαΐου θα γίνει ψηφοφορία. Η ψηφοφορία στη 15-16 Ιουνίου στους προϋπολογισμούς και τον Ιούλιο θα πάει στην Ολομέλεια. Αυτά και παρακαλώ τον συνάδελφο Λεβαντόφσκι, αν επιθυμεί, να προσθέσει κάτι. Δεν γνωστό το χρονοδιάγραμμα. Ήμασταν πιο γρήγοροι από την Κομισιόν αυτή τη φορά. Η Κομισιόν περιμένει το Βρετανικό δημοψήφισμα. Γι' αυτό δεν κάνει την αναθεώρηση πριν το, πριν το δημοψήφισμα των Βρετανών. Μάλλον μετά τον Ιούνιο θα προβεί στην αναθεώρηση. Εγώ είμαι ανοιχτό σε διάλογο. Αυτό που έχει σημασία είναι να εσωματώσουμε τι δικέ μα προτεραιότητε. Γιατί συμφωνήθηκαν ομόφωνα. Ό,τι και να συμβεί, και συμβαίνουν πάρα πολλά, έτσι, και για το ΕΦΣΙ και παντού, δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος των ομοφώνων συμφωνηθέντων πραγμάτων. Χρειαζόμαστε να προχωρήσουμε, είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Μπορώ να συνομιλήσω και με τις άλλες ομάδες, ούτω ώστε σε επίπεδο ίδρυ τουλάχιστον να εκφραστούμε με μία φωνή, ομόφωνα. Έχουμε ξεκάθαρες προτεραιότητες, πρέπει να τις περασπιστούμε, τις συμφωνήσαμε και νέες ανάγκες, νέες προκλήσεις πάντα θα πρέπει να αναγνωριστούν, αλλά όχι εις βάρος των δικών μας προτεραιοτήτων. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Και πάμε στο επόμενο θέμα, αποστολή αντιπροσωπεία στη Ήθρα στη Λουμπλιάνα. Προβλέπεται ενημέρωση. Ο συνάδελφος Κόφορτ θα μας ε, κάνει μια σύντομη ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια αποστολή. Ήταν μια αποστολή διήμερη επισκεφθήκαμε την Αίζα αλλά και άλλα μέρη εντός και εκτός Λουμπλιάνα. Δεν είναι και πολύ συναλφοί εδώ σήμερα αλλά είναι πολύ σημαντικό να σας ενημερώσουμε. Ο κ. Ρούμπικ ήταν επίσης μέλος της αποστολής οπότε θα μπορούσε να με συμπληρώσει. Την Πέμπτη αφιερώσαμε την με τη μέρα στην επίσκεψη της ΕΙΖΑ να σας ε, πω ποια ήταν τα ενδιαφέροντα σημεία. Ε, η ΕΙΣΑ έχει συνεργαστεί με την Ήτρα ε, στο παρελθόν πολύ αποδοτικά και χαίρομαι που καταφέραμε και επισκεφθήκαμε το, τα κεντρικά της γραφεία, ε, είδαμε και τους εργαζόμενους, όχι μόνο τα διευθυντικά στελέχη. Καταρχήν μιλήσαμε για τους κωδικούς ε, ε, δικτύων και το πώς εφαρμόζονται στα δίκτυα ε, φυσικού αερίου. Έχουν γίνει πολλά πράγματα, θα πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα όμως. Το ίδιο και για τα ηλεκτρικά δίκτυα. Τα εικόδικες θα πρέπει να ε, εφαρμοστούν και με τρόπο μάλιστα ομοιόμορφο. Μετά συζητήσαμε για τις ε, βασικές προκλήσεις της Ενεργειακής Ένωσης και της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς. Εξετάσαμε την έκθεση παρακολούθηση των αγορών της ΕΙΖΑ. Ε, είναι πολύ χρήσιμη αυτή η έκθεση. Να υπογραμμίσω τα εξή. Η τάση είναι μείωση των τιμών σε όλες τις αγορές, χωρίς αυτό όμως ε, να ε, βλέπουμε να αντικατοπτρίζεται και στις τιμές καταναλωτού. Είναι κρίμα οι καταναλωτές ε, να μην αγοράζουν σε φτηνότερες τιμές τα προϊόντα τα οποία παράγονται σε, με χαμηλότερο κόστος ενέργειας. Η έκθεση επίσης της ΣΕΙΖΑ αναφέρει ότι, σχετί, ε, ότι βασίζεται στα κράτη-μέλη να παράσχουν στατιστικά στοιχεία σε εθελοντική βάση και αυτό βέβαια δημιουργεί μερικές φορές προβλήματα στη σύγκριση και στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Οπότε ο διευθυντής ζήτησε περισσότερες εξουσίες σε αυτό το θέμα. Θα πρέπει εμείς να δούμε πώς εφαρμόζεται η, ενεργειακή, η εσωτερική ε, ενεργειακή ένωση. Επίσης μιλήσαμε και για συγκεκριμένα προβλήματα στο εσωτερικό κρατών μελών αλλά και διασυνοριακά. Μιλούμε για εμπόδια, υλικά εμπόδια αλλά και άειλα Μιλούμε για έλλειψη υποδομών, για διαφορές όμως και όμως για δια, κανονιστικές διαφορές. Ε, μονάδες διασύνδεσης οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς κάτι που οδηγεί σε στρεβλώσεις κλπ. Στην τρίτη σύνοδο μιλήσαμε για το πακέτο ε, Ενεργειακής Ένωσης και για μελλοντικές βελτιώσεις. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Θα πρέπει όλα όμως να βασίζονται σε αναλύσεις κόστους κόστους-οφέλους ε, και να μην γίνονται πρόχειρα. Μετά, ένα σημαντικό θέμα συζήτηση ήταν η παρουσίαση και συζήτηση για τη ενεργειακή ένωση σε σχέση με το μελλοντικό ρόλο της ΕΙΣΑ και τις δραστηριότητές της. Όπως γνωρίζετε, περιμένουμε η Κομισιόν μέσα στο 2016 να προτείνει ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΖΑ ε, στο πλαίσιο αυτό θα συζητηθούν οι σημερινές αρμοδιότητες, οι μελλοντικές αρμοδιότητες και τα μέσα που θα διαθέτει, οι πόροι που θα διαθέτει. Είναι μια συζήτηση που έχει γίνει πολύ και στο παρελθόν. Θα πρέπει να ε, ενισχυθεί η ΑΙΖΑ, γιατί αλλιώς ε, δεν μπορεί να επιτελέσει το ρόλο της. Σε ό,τι διαφορά το θέμα της ε, ε της ε, ε, χονδρικής αγοράς ενέργειας, ε, με πολύ ενδιαφέρον είδαμε ότι η ΕΙΖΑ παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την αγορά αλλά και πάλι μας υπογράμμισαν ότι θα πρέπει η παρακολούθηση αυτή να γίνεται με όνομα 26 άτομα προσωπικό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η αντίστοιχη ε, επιτροπή ε, έχει 89 άτομα προσωπικό. Καταλαβαίνετε τη διαφορά μεγέθους. Η συζήτηση έκλεισε με συγκεκριμένε παρατηρήσει από εμά και από το Διευθυντή. Στηρίζουμε την ΕΙΣΑ, είναι ένα τα συμπεράσματα. Εξακολουθούμε να προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε παρκή πόρου και δυναμικό. Και σίγουρα χρειάζεται να συνεργαστούμε περισσότερο στο μέλλον θα λάβει χώρα ε, μια συνάντηση της ε, αντίστοιχης ε, ομάδας της Ίτρε με την ΕΙΣΑ και τέλος να πω το εξής επισκεφθήκαμε το Ινστιτούτο Ιώζεφ Στέφαν στη Λουμπλιάνα είναι λίγο εκτός Λουμπλιάνας, εκτός πόλης είναι ένα ε, ε οργανισμ, ο ερευνητικός οργανισμός της Σλοβενίας ασχολείται με βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία. 960 άτομα προσωπικό ε, που ερευνούν στη φυσική, τη χημεία, βιοχημεία, ηλεκτρονική, ε, ενέργεια, ε, χρησιμοποίηση ενέργειας, περιβαλλοντικές επιστήμες, ε, τεχνολογία πληροφορίας κλπ. Το ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης κατατάσσει αυτό το Ινστιτούτο μέσα στα καλύτερα της Ευρώπης. Συζητήσαμε επίσης ε, για τεχνολογίες ε, σχάσης και σύνδεξης. Δεν θα σας πω πολλά πράγματα όμως γι' αυτό. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη. Νομίζω ότι μιλώ εκ μέρους ε, όλων ε, λέγοντα ότι ήταν πολύ χρήσιμη και θα πρέπει να συνεχιστεί και στο μέλλον αυτή η επαφή, ιδιαίτερα με την ΕΙΖΑ. Ευχαριστούμε πολύ και για μένα ήταν εντυπωσιακό το ταξίδι γιατί εκεί διαμορφώνεται το μέλλον της Ευρώπης. Δεν είναι εύκολο 28 ρυθμιστικοί ε, φορείς να συντονιστούν σε ευρωπαϊκό πλαίσιο γιατί η παράδοση ήταν διαφορετική. Ο καθένας ήταν υπεύθυνο για κάθε κράτος. Και τώρα υπάρχουν ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριότητες. Χρειάζεται λοιπόν και άλλη δράση εδώ, ώστε οι αντιλήψεις για την κοινή αγορά να ε, ε, συντονιστούν και με τους εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς ώστε να μην υπάρχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, αλλά να υπάρχει συνέργεια. Γι' αυτό... Καλέσαμε και μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ε, στη χώρα, ούτως ώστε να συνεργαστούμε και να δώσουμε ε, μια όθηση. μπορούμε να ε, υπερβούμε τα εθνικά σύνορα σε αυτούς τους τομείς και να μην δημιουργήσουμε καινούρια. Δεν θέλουμε στα εθνικά ε, δεν θέλουμε ε, επαναφορά των εθνικών συνόρων. Καλό είναι να φέρουμε κοντά τις περιφέρειες της Ευρώπης που εκπροσωπούνται και στην Επιτροπή των Περιφερειών και πρέπει να συνεργάζονται. Όλα αυτά στην πράξη δεν είναι εύκολα, αλλά ε, θα πρέπει οι παραμεθόριες περιοχές να συνεργάζονται και να δοθεί σε αυτές προτεραιότητα. Έτσι θα προχωρήσουμε ήδη. Υπάρχει ανάθεση μιας μελέτης σχετικά με τις ικανότητες. Θα ολοκληρωθεί το 17 και θα δούμε τι θα βγει και από εκεί. Και όπως είπα, οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς πρέπει να αναλάβουν δράση. Ιδιαίτερα στη Γερμανία βλέπουμε ότι ε, δεν μπορούν να λυθούν τα προβλήματα μόνο σε επίπεδο εθνικό. Οπότε θα πρέπει να απασχολήσουν τα προβλήματα της κάθε χώρας και της άλλες χώρες, όχι μόνο τις γειτονικέ. Μιλάμε για ένα εγχείρημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που ανοίγει και πολλές ευκαιρίες. Θα πρέπει να δούμε τη στρατηγική πρόκληση που υπάρχει. Ε, για την αιωλική ενέργεια ή την ηλιακή ενέργεια και εδώ θα πρέπει να συνεργάζονται οι περιφέρειες ε, στη... παντού, στη Δύση, Ανατολή, Βορρά, Νότο. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας του συνδυασμού που μπορούμε να κάνουμε για προσφορά ηλιακής ενέργειας, γεωθερμικής ενέργειας, ολικής ε, ενέργειας. Όλα αυτά θα τα ε, λάβουμε υπόψη μας αν θέσουμε υπό έλεγχο τα βασικά προβλήματα της κλιματικής αλλαγής. Είναι ε, πολύ ενδιαφέρουσα και η συνεργασία με το ΜΠΕΡ και την Ευρωπαϊκή Διαστημική ε, ε, Ευρωπαϊκό Διαστημικό Οργανισμό, ε, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, διότι υπάρχουν στην τεχνολογία σημεία επαφής που μπορούμε να τα ε, αξιοποιούμε. Υπάρχει συνεργασία BEREC και ε, υπάρχουν επίσης οι ευφυείς μετρητές. Όλα αυτά είναι ζητήματα που δεν μπορούμε να τα βλέπουμε μεμονωμένα μόνο σε ένα κλάδο. Άρα θα υπάρχουν συνέργειες, συνεργασίες και γι' αυτό είναι σημαντικό η, τόσο σημαντική η ΑΕΣΑ. Οι προτεραιότητές της μας βρίσκουν σύμφωνους και θα πρέπει να δούμε και τι νομοθετικά πλαίσια χρειάζονται ακόμη. Σύντομα θα γίνει μια μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα εδώ στο Κοινοβούλιο. Με αυτό το ταξίδι ελπίζω ότι μπορέσαμε να δείξουμε ότι επί τόπου γίνεται εντατική δουλειά. Εγώ αποκόμισα πολύ θετικές εντυπώσεις. Αυτό που χρειαζόμαστε και το είδαμε επιτόπου είναι ότι χρειάζεται μια αξιολόγηση των ε, βασικών ε, στρατηγικών. Ε, είδαμε επιτόπου το ΜΕΡΕΚ, την ΕΙΣΑ, υπάρχει επιτροπή. Θα πρέπει όμως να βελτιωθούν οι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ αυτών και η επιτήρηση της αγοράς ε, που γίνεται στην ε, Λουμπλιάνα θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και αλλού. Ε, θα πρέπει δηλαδή να δούμε πώς ρέει στην πραγματικότητα η ενέργεια στην οικονομία, πώς ενέργεια και οικονομία συνδυάζονται. Είναι πολύ σημαντικό ότι η ηλεκτρική ενέργεια ε, ε, λειτουργεί και με βάζει φυσικές ιδιότητες ε, και όχι μόνο οικονομικές. Τώρα και με το σύστημα, τα συστήματά μας IT προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες σύνδεσης και ο κύριος Βόλτερ μίλησε για αυτά τα θέματα νωρίτερα. Ε, ενδεχομένως ε, τα έσοδα από το, την εμπορία των ε, εκπομπών ε, μπορούμε να την αξιοποιήσουμε στα δίκτυα, επενδύοντας στα δίκτυα. Τα μέσα που θα αποκτήσουμε από το διοξίδιο ε, του άνθρακα και τον πληστηριασμό που θα γίνει εκεί μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε πολλά έργα. Η ενεργειακή οικονομία χρειάζεται νέες δομές ώστε τους ε, στόχους μας να τους ε, συνδυάσουμε και με το γενικότερο στόχο του 30%. Η επίσκεψη στη Λουμπλιάνα προώθησε όλους αυτούς τους προβληματισμούς. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Γραμματεία, τον Έρνες την Ιβάνα που μας συνόδευσαν και φρόντισαν για την ε, άψογη διεξαγωγή της επίσκεψης. Εμείς χρειαζόμαστε την επαφή με τους ενδιαφερομένους και αυτός είναι ο στόχος μας να διατηρήσουμε την επαφή μας. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις Θέλω να ευχαριστήσω όλους. Ε, η διακόπτη συνεδρίαση και θα συνεχιστεί σήμερα το απόγευμα σε αυτή την αίθουσα στις 3. Λύεται η συνεδρίαση.